έρθει αργότερα και με την... Ε, εμείς, εγώ θα προεδρεύσω τη συνεδρίαση. Ε, ήθελα να πω ότι υπάρχουν ορισμένες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Θα ξεκινήσουμε με τις ανακοινώσεις Προέδρου. Μετά θα περάσουμε στο 5 δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στι διεθνείς Εμπορικέ Συμφωνίε θα ακολουθήσουν τι ανακοινώσει του Προέδρου, θα είναι δηλαδή το σημείο 3 της ημερήσιας διάταξη. και μετά θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη, γυναίκα, με, τη βία κατά των γυναικών σε ένοπλε συγκρούσει και μετά θα περάσουμε ε, στην, ε, στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των ε, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν αντιρρήσεις, αν όχι μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ρίτσαρντ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ημερήσια διάταξη, μόνο για τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Είχα ζητήσει από τη Γραμματεία ένα έγγραφο εγγρασίας για το οποίο η κυρία Χάουταλα είχε πει ότι είναι προτεραιότητα για τον Ιανουάριο. Είμαστε ήδη στο Μάρτιο. Είμαι σίγουρος ότι έχει δρομολογηθεί η επεξεργασία του, αλλά θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται γιατί για μένα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα Μιλάω για την υπηρεσία, την εξωτερική ε, υπηρεσία, την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Είναι κάτι το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα και θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Μικρόφωνο παρακαλώ. Κοιτάξτε, στο Στρασβούργο θα το συζητήσουμε. Το σημείωμα της γραμματείας θα συζητηθεί στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις? Ωραία, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Πολύ ωραία. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Το δεύτερο θέμα είναι οι ανακοινώσει της Προέδρου. Πρώτον, για τον Ρολάντο Ζαπάτα Ταμάιο, τον ε, κουβανό πολιτικό ε, φυλακισμένο, πέθανε στις 24 Φεβρουαρίου μετά από απεργία πείνας. Ε, σε μια καταστολή συνελήφθη μιας μεγάλης εξέγερσης στην Κούβα. Πρόκειται για ε, το λόγο για τον οποίο ο Σφάλτο Φάγια πήρε το βραβείο Ζαχάροφ το 2002. Ο Ορλάντο Ζαπάτα Ταμάιο ε, καταδικάστηκε το Μάιο του 2004 σε τρία χρόνια φυλάκιση. Στη συνέχεια ε, πέρασε, ε, αποδίκη πολλές φορές ε, για ανυπακοή και ε, υποκίνηση σε εξεργέρσεις. τελευταία φορά 2009, 36 χρόνια ε, ήταν αγωνιστής και η τελευταία του απεργία πείνας είχε σκοπό να, ε, να αντιταχθεί στις κακές συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές. Πολλές φορές ζητήσαμε την άνεφορον ε, απελευθέρωση όλων των πολιτικών ε, κρατούντων ε, στην Κούβα. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε μία πρόταση στην Ολομέλειά μας στο Στρασβούργο να γίνει μία συζήτηση με ψήφισμα σε σχέση με την Κούβα. Μπορώ να ζητήσω την υποστήριξή σας ε, για συζήτηση με ψήφισμα στην Ολομέλεια του Στρασβούργου την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη ανακοίνωση για την 54η Σύνοδο. Διακόπτη Πρόεδρος. Με την 54η Σύνοδος της ε, Διάσκεψης για την Κατάσταση των Γυναικών στο Πεκίνο, 15 ε, συν, από ό,τι καταλαβαίνω από το έγγραφο, η Χάιντι Χάουταλα μετέβει στην 54η Σύνοδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες και επειδή πολλά από τα ζητήματα είχαν άμεση σχέση με τις γυναίκες στις ειρηνευτικές, στην ειρηνευτική διαδικασία. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, αλλά όταν θα έρθει η κυρία Χάουτελα, η πρόεδρός μας, αν έχετε ερωτήσει σε σχέση με το θέμα αυτό, θα ε, απαντήσει με χαρά. Επίσης, ε, η κυρία Χάουταλα ήταν τμήμα της αντιπροσωπείας ε, της εξεταστικής στην Λευκορωσία την περασμένη εβδομάδα. Επικεφαλής ήταν ο Κρίστιαν Βικένεν. Από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου ο σκοπός ήταν ε, να ε, εξεταστεί το ενδεχόμενο της ε, Λευκορωσίας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΟΗΕ, όπως επίσης και τα ζητήματα της, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, όπως επίσης και τα ζητήματα των εθνικών μειονοτήτων στη Λευκορωσία. ψήφισμα για τη Λευκορωσία σύμφωνα κατόπιν ε, της ε, ε, για την, την έκθεση της έκθεσης για τις μειονότητες στην Λευκορωσία θα υπάρξει στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Yes, so those are all announcements. Αυτές ήταν οι, ανακοινώσει ανακοινώσεις της Προέδρου, συγγνώμη, για σήμερα. Και τώρα νομίζω μπορούμε να περάσουμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που όπως είπα προηγουμένως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές ε, συμφωνίες. David Μάρτιν, ο συντάκτης γνωμοδότησής μας. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Ντέιβιν Μάρτιν, που είναι ο συντάκτης του νομοδότησης, και τον Γκρεκουάρ Τερί, ο οποίος επίσης θα παρέμβει για το θέμα αυτό, και εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ε, θα φτάσει σε λίγο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον David Μάρτιν. Ευχαριστώ και καλημέρα. Έχει μεγαλύτερη ευκαιρία τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επηρεάσει το περιεχόμενο των εμπορικών συμφωνιών από ότι το παρελθόν λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας. Είμαστε τώρα ισότιμοι εταίροι στην έγκριση εμπορικών συμφωνιών με το Συμβούλιο Υπουργών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε για να πούμε το ναι ή το όχι το τέλος της διαδικασίας. Θα πρέπει να αρχίζουμε να εμπλεκόμεθα από την αρχή της διαδικασίας, να παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις, να πούμε ναι ή όχι όταν θα έρθει το θέμα της έγκρισης και μετά να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε για να ε, βεβαιωνόμαστε ότι ε, τηρούνται οι αρχές επί των οποίων βασίζονται οι συμφωνίες. Και αυτό ε, απασχολεί ιδιαίτερα και την παρούσα υποεπιτροπή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι θέματα βέβαια και διεθνού δικαίου και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οφείλει να φροντίζει και αυτό να παρακολουθεί ότι οι αναμειγνιόμενες συμβαλόμενες χώρες ψεύονται τις ελίτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και συμφωνίες με GSP Plus να έχουν ρήτρε για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη εργασία κτλ. Και ο στόχο της νομοδότησής μας είναι να εξετάσουμε με ποιον τρόπο μπορούν να επιβάλλονται καλύτερα, μπορείτε, μπορεί να επιβάλλεται καλύτερα η τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσω εμπορικών συμφωνιών. Πρώτον, τα οριζόντια θέματα. Προφανώ εδώ τίθεται θέμα GSP συν για να επωφεληθούν από την GSP syn πρέπει ε, να βασιστούμε σε ορισμένες βασικές συμβάσεις ε, του Διεθνούς, Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας περιβαλλοντικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εάν δεν τηρούνται οι προδιαγραφές αυτές, τότε τα πλονεκτήματα της GSP μπορούν να αποσυρθούν. Για πολλές από τις αναπτυσσόμενες χώρες αυτές είναι σημαντικές. Σε αυτά είναι σημαντικά πλονεκτήματα. Μείωση δασμών, εξακολουθούν οι όροι της GSP να προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες που συμβάλλονται σε εμπορικές συμφωνίες. Υπάρχει όμως μια έλλειψη συνέχειας στο ποιος λαμβάνει τα πλεονεκτήματα, τα ευεργετήματα της GSP+. Στο τελευταίο γύρο, ίσως και δικαίως αποκλείσαμε το Πακιστάν από το GSPC με στην βάση του ότι δεν τηρούσε πολλές από τις προδιαγραφές ε, του ILO πάλι βασισμένοι στις ίδιες παραμέτρους ίσως καλώς αποκλείσαμε το Πακιστάν όμως ορισμένες άλλες χώρες περιλήφθηκαν και διότι κανείς ποια είναι εν τέλει τα κριτήρια. Διότι αν τα κριτήρια είναι περισσότερο μια real politik, το Πακιστάν είναι μια χώρα που θέλουμε να συμβάλλουμε στην σταθεροποίησή της. και χώρες οι οποίες ε, εν τέλει εντάσσονται στην GSV Plus Πάλι σωστά νομίζω αποφασίσαμε να αποκλείσουμε την Σρι από τα ευεργετήματα της gsp λόγω της κατάστασης ανθρώπινων δικαιωμάτων εκεί, αλλά δεν αρνούμεθα να αρχίσουμε έστω μια έρευνα στην Κολομβία. Στην Κολομβία όπου ...60% των φόνων συνδικαλιστών γίνονται στην Κολομβία. Για μόνο το λόγο ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν συνδικαλιστές. Ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν στην Κολομβία. Δεν κάνουμε τίποτα εκεί, αν από την άλλη μεριά κινούμαστε για να αποκλείσουμε τη Σρι Λάνκα. Υπάρχει μια έλλειψη συνεχτικότητα. Όταν το συζήτησα αυτό με αξιωματούχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φάνηκε το μέτρο να μην είναι τόσο πολύ εάν η συγκεκριμένη χώρα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι δεσμεύσει της σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας και η ερμηνεία πάντως που δίνω στις εξηγήσει τους είναι εάν θα έπρεπε να δείχνει κάποια τάση να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα δίνοντας τότε τα ευεργετήματα της DSPC και τα λοιπά την ενισχύουμε υποτίθεται σε αυτήν την πορεία. Περισσότερο λοιπόν είναι μια ερμηνεία του τι θα συμβεί εάν δοθούν ή αν αφαιρεθούν τα ευεργετήματα αυτά. Ίσως φαίνεται λογική αυτή η προσέγγιση, αλλά δεν έχει καμία ε, συγκεκριμένη βάση ποιε βελτιώσει πρέπει να υπάρχουν, ποια είναι τα benchmarks για τι βελτιώσει αυτέ. Και εν τέλει νομίζω ότι απλώ είναι η εικόνα που έχει ο καθενό και εν τέλει μα αρέσει ή δεν μα αρέσει η χώρα. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά αυτό βέβαια δεν αποτελεί ικανοποιητική βάση για να ασκηθεί πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εξήγηση που δόθηκε για την Κολομβία, για, το τι δεν γίνεται, για, για, ποιο λόγο δεν γίνεται δηλαδή εκεί έρευνα, είναι διότι η Κομισιόν θεωρεί ότι η ενασχόληση με την Κολομβία τους ενισχύει στην πορεία προς ε, μια βελτίωση ενώ το αντίθετο συμβαίνει στην Σρι Λάνκα. Αλλά αυτά βασίζονται περισσότερο στην εικόνα που έχει ο κάθε αξιωματούχο για ε, την ε, συγκεκριμένη χώρα και δεν, έχει, δεν βασίζεται σε εμπειρικά ή άλλα αντικειμενικά στοιχεία. Πάλι αναφέρομαι στην Κομισιόν και καταλαβαίνω βέβαια τις δυσκολίες της δουλειάς τους, τα κριτήρια των επενδύσεων πιο διστακτική να αναπτυχθούν. Αν όμως κάνουν μια πρόταση για αφαίρεση ενός ευεργετήματος, δεν είναι βέβαιο ότι θα περάσει από το Συμβούλιο, του Συμβουλίου Υπουργών. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε συχνά είναι να γίνονται συζητήσεις και κλεισμένων των θυρών, συζητήσεις μεταξύ κομισιών και υπουργών ή του είπα του με την έννοια δηλαδή, εάν κάνουμε αυτή την πρόταση θα την υποστηρίξετε στην περίπτωση της Κολομβίας είναι προφανές ότι το Συμβούλιο δεν πρόκειται να δεχθεί να άρει τα ευεργετήματα της GSPC. Η δική μου γνώμη είναι ότι ποτέ δεν θα είναι ξεκάθαρα άσπρα ή μαύρα τα πράγματα. Βεβαίω πάντοτε πρέπει να προσπαθούμε να καθιερώσουμε ένα ξεκάθαρο σύνολο κριτηρίων για το εάν μια χώρα ενδείκνεται να ευεργετηθεί από το GSP ή όχι. Υπάρχουν βέβαια και άλλε περιοχέ με τι οποίε κάνουμε, διεξάγουμε εμπόριο από τι χώρε που προηγουμένω. Τώρα, η άλλη, ο άλλο χώρο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών στι διαπραγματεύσει με τρίτη χώρα για τέτοια συμφωνία έχουμε πάλι ε, ε, ε, ρήτρε σχετικά με το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εργασία ώστε να οθούνται οι χώρες να βελτιώνουν την κατάσταση σε αυτά. Κορέα για παράδειγμα για να υπογράψουν συμβάσεις του ILO που μέχρι τώρα τις στέκονταν, δεν τις υπέγραφαν για να έχουν τελικά, να, να μπορέσουν να υπογράψουν μια συμφωνία εμπορίου μαζί μας. Βέβαια, Αυτή τη στιγμή υπογραφεί η συμφωνία, οι προσπάθειες αυτές εξαφανίζονται, διότι για να αρθεί μια συμφωνία χρειάζεται ξανά πρόταση κομισιών κτλ. Αρχίζουν λοιπόν να επενδύονται πάρα πολλά συμφέροντα στην συμφωνία αφού ευεργετούνται πολλές περιοχές, χώρες και ούτω καθεξής και από ό,τι ξέρω ποτέ δεν ήρθε κάποια συμφωνία κάποια εμπορική συμφωνία. Ορισμένες φορές ήρθησαν τα ευεργετήματα της GSP ακόμα και με το Ισραήλ, όπου θα υπήρχε δικαιολογία, ούτε καν προτάθηκε να έρθει η συμφωνία. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω κατά πόσον είναι εφικτό, στο μέλλον και θα ήθελα το Κοινοβούλιο εκεί να πιέσει να, να γίνει πιο εύκολο, ας το πω καλύτερα έτσι, να εφαρμόζονται οι αρχές ανθρώπινων δικαιωμάτων είτε στη βάση της ομοφωνίας, είτε δίνοντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα πρωτοβουλίας να άρει ή να αναστείλει μια συμφωνία και το κατεξής. Θα ήθελα το Κοινοβούλιο να έχει ένα ξεκάθαρο ρόλο σε ό,τι αφορά την υποβολή προτάσεων για την αναστολή μιας ε, συμφωνίας εμπορίου ε, ελεύθερων συναλλαγών δηλαδή. Αυτό δεν θα λύσει τα προβλήματα των υφιστάμενων FTAs, αλλά μπορεί ωστόσο να βελτιώσει τα πράγματα για το μέλλον, για μελλοντικές συμφωνίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάρτιν. Έχουμε ανταλλαγή απόψε, αλλά δεν έχουμε έγγραφο Αλλά στα έγγραφά σας έχετε ένα έγγραφο από την ε, Διεθνή Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Γκρεγουάρ Τερή ε, εκπροσωπεί την ε, Διεθνή αυτή Ομοσπονδία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Στα γαλλικά θα μιλήσω. Καταρχά, ευχαριστώ πολύ την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μα προσκάλεσε στο πλαίσιο τη ανταλλαγή απόψεων, η οποία είναι βέβαια πολύ πρόημη, γιατί όπω είπατε και εσεί, δεν υπάρχει κείμενο επί του οποίου να δουλέψουμε. Για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε εδώ, γιατί η οργάνωσή μα εδώ και πολλά χρόνια έχει ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό της, ε, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των ε, ε, εμπορικών ε, συμφωνιών και των διεθνών συμφωνιών. Είναι ένας, ένα ζήτημα που μας απασχολεί πολύ περισσότερο για πολλούς λόγους που είναι σημαντικό να τους συζητήσουμε. Πρώτον, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλές φορές, ε, έχει πολλαπλασιάσει πλέον ε, τις εμπορικές της διαπραγματεύσεις και τις εμπορικές της συμφωνίες με τρίτες χώρες. Δεν μπορούμε λοιπόν να παραγνωρίζουμε τη σημασία αυτών των διαπραγματεύσεων των εμπορικών που πραγματοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια. Εδώ σημαντικό πλαίσιο στα πλαίσια της όλης εξέλιξης με την ε, ε, επικύρωση της συνθήκης της Σαββόνα το άρθρο 218 της συνθήκης αλλά και η νέα διαθεσμική συμφωνία ε, προχωρεί, μάλλον ε, δίδει μια αρμοδιότητα ιδιαίτερη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο που παρακολουθεί τις διαπραγματεύσει σε κάθε φάση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο μπορεί να παρέμβει σε οποιαδήποτε φάση και όχι έτσι στενά όπως λέγαμε παλιά και απλά και μόνο λέει ναι ή όχι όπως είπε και ο συγητής. λοιπόν αυτή η προοπτική είναι ιδιαίτερα ενεργητική, ενεργή υπάρχει δραστήρια, το πούμε έτσι. Και υπάρχει μια αναγνώριση ιδιαίτερη τη σημασίας στο διεθνέ κοινωνικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών. Αναφέρω επίση τον ε, διευθυντή ε, του ΠΟΛ που είπε σε μια πολύ σημαντική δήλωση ο Πασκάλ Λαμί είπε τον Ιούνιο ότι το άνοιγμα παρομοίων συμφωνιών και η συμπερίληψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι κάτι το αυτόνομο. Χρειάζονται ρυθμίσει γενικέ και δίκε και αναρτιούνται οι νομικοί εάν ε, ο ΠΟΕ ακριβώ σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά είναι σαφή θετική απάντηση. Έχουν τη θέση του πάνω απ' όλα στο διεθνέ δίκαιο γιατί ακριβώ επιβάλλονται. Εδώ στην παρουσίαση τη σύντομη μου θα ήθελα να ξεκινήσω από το σημείο αυτό να σας πω ξεκινώντας ε, για το διεθνές δίκαιο ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα σε εμπορικές συμφωνίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα ακριβώ, ε, κάτι που θα πρέπει να είναι αυτόματο χωρί καμία συζήτηση και σε περισσότερα πολιτικά θέματα στα πλαίσια της εξωτερική πολιτικής Ευρωπαϊκή Ένωση, στι ιδιαίτερε προσπάθειε ώστε αυτή η εξωτερική πολιτική να κρίνεται από συνοχή σε όλου του τομεί, ποια είναι η θέση τη συνοχή και ορισμένων προποθέσεων. Πρώτο σημείο στο διεθνέ δίκαιο και γι' αυτό ακριβώ ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει θεωρητική συζήτηση πάνω σε αυτό. Τα κράτη-μέλη αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, νομικά ε, είναι υποχρέα λόγω διεθνών υποχρεωσών τους ε, για τα δικαιώματα και τα κοινωνικά οικονομικά δικαιώματα και αυτή η Διεθνή Συμφωνία για τα κοινωνικά οικονομικά δικαιώματα συμπεριλαμβάνει και μια υποχρέωση μια συνεργασία, μια διεθνή αρρωγή. Και το άρθρο 2.1 και το άρθρο 11 λένε ακριβώ ότι οι υποχρεώσει αυτέ συνεπάγονται ότι δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στι τέτοιε χώρε. Η Επιτροπή ακριβώ ανέπτυξε την έννοια αυτή και μας εξηγεί ότι στα κράτη-μέλη των ΗΕ Εθνών εκεί υπάρχει υποχρέωση να ελέγχουν ότι όλες οι διεθνείς συμφωνίες τις οποίες διαπραγματεύονται και κλείνουν μέτρητες χώρες δεν προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί αλλά αντίθετα βοηθούν για το σεβασμό αυτών η υποχρέωση διεθνή στα πλαίσια όλων των διεθνών συμφωνιών και εμπορικών είναι πρόφανης ε, τα κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι μέσω των συμφωνιών αυτών δεν προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες. Ε, και γνωρίζουμε σήμερα, ε, άλλωστε υπάρχουν και αποδείξεις, ότι οι εμπορικές συμφωνίες, αυτό αποδείχθηκε στα Ηνωμένα Έθνη και ο κ. Λαμί το αναγνωρίζει, ότι μπορεί να υπάρχει σαν αποτέλεσμα κάτι το θετικό αλλά και κάτι το αρνητικό όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτη χώρα. Σήμερα τι μας ενδιαφέρει και πριν από δύο χρόνια ε, δημοσιεύθηκε άλλωστε να δούμε τα μέσα τα πραγματικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να δούμε ότι πραγματικά σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων και να βεβαιωθούμε αν υπάρχει θετικός ή αρνητικός αντίκτυπος και αν είναι κάτι το αρνητικό τότε να αλλάξουμε τους όρους συμφωνίας αυτής τι διαπιστώνουμε, ότι δεν έχει κανένα μέσο η Ευρωπαϊκή Ένωση από διαφορετικής πλευράς, θεσμικής πλευράς να αποδείξει ότι θα έχουν μια θετική, ένα θετικό αντίκτυπο και όχι αρνητικό αυτές οι συμφωνίες. Τώρα όμως έχουμε το ένα μέσο που επιτρέπει να δω, από πριν τον αντίκτυπο στην αηφόρο ανάπτυξη, αλλά ε, όχι όμως ειδικό μέσο ότι δεν θα υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω να προσθέσουμε κάτι εδώ και αυτό είναι το κύριο σημείο, θα είμαι σύντομος. Είναι η σημασία το πώς το μέσο αυτό, το εργαλείο να το αναπτύξουμε σε διαθεσμικό επίπεδο, το human rights ε, κλπ ε, και το οποίο θα μπορούσε να είναι, δεν είμαστε αντίθετοι, θα μπορούσε να αποτελέσει μια διεύρυνση του όρου αναφοράς του Sustainable Impact Assessment. Ε, δεν πρέπει να είναι μόνο ένα καινούριο εργαλείο, ίσως η αναφορά να είναι περισσότερο ευρεία και να μπορέσουμε έτσι να είμαστε σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τις υποχρεώσεις της σε διεθνές επίπεδο. Να δούμε το, το δεύτερο σημείο, πέρα από το διεθνές δίκαιο, περισσότερο πολιτικό είναι, αλλά ειδικά ενδιαφέρον στα πλαίσια της νέας συνθήκης της Αβώνας. Ε, θέμα συνοχής και ορισμένε προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις ε, είναι κάπως ε, ταμπού σαν όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Επαφέ μα με υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι όμω αυτή οι υποθέσεις μια πραγματικότητα τη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή. Ένωση. Ε, το συν βασίζεται σε αυτέ τι προποθέσει ε, θετικέ. Η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε συμφωνία από το 95 που κλείνω με τρίτες χώρες ε, συνεπάγεται και κάτι σχετικά με αυτές τις προϋποθέσεις από τη στιγμή που εγγυόμεθα στο άρθρο 2 συμφωνίες αυτές ε, τα βασικά στοιχεία είμαστε σε πλαίσια διεθνούς δικαίου σε αυτή την δυνατότητα παγώματος συμφωνίας εάν τα κριτήρια, τα σημαντικά αυτά σημεία που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι δημοκρατικές αρχές αν δεν γίνονται σεβαστά αυτά Υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις λοιπόν και εφαρμόζονται κυρίως στα πλαίσια της Συμφωνίας του Κοτονού. Βλέπουμε de facto ακριβώς σε περίπτωση που δεν υπάρχει πια δημοκρατία, σε περίπτωση πραξικοπήματος ακόμα, το 96 άρθρο χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση της Συμφωνίας του Κοτονού για να παγώσει τη συμφωνία αυτή. Για μας αυτό που έχει σημασία είναι αυτές οι προϋποθέσεις ε, για τη χρήση της ρήτρα αυτής ε, και μιας έρευνας παρόμοιας ε, και αυτών των των θετικών σημείων, αν αυτά συζητούνται, να συζητούνται σε θεσμικό επίπεδο για περισσότερο συνοχή στην εφαρμογή τους. Και σημαντική προοπτική με την νέα συνθήκη της Σαββόνας, με το άρθρο 21. Το άρθρο 21 λέει σαφώς ότι απαιτείται ιδιαίτερη συνοχή στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε τομέα ξεχωριστά και επίσης ε, υπάρχει ανάγκη για το mainstreaming ε, βασικών ε, θεμελιδών δικαιωμάτων, τα ανθρώπινα δικαιώματα ας πούμε, στο πλαίσιο όλων των πολιτικών και σε κάθε τομέα της εξωτερικής πολιτικής αυτό που θέλουμε και είμαστε μια προκαταρτική φώση, δεν έχουμε ακόμα κάτι που να έχει αποφασιστεί, αλλά επιθυμούμε το δημόσια σε διαθεσμικό επίπεδο να γίνει μια συζήτηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να βοηθήσει και να ασχοληθεί με το θέμα για να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θετήσει μια πολιτική με συνοχή, όχι με δύο στάνταρντ, αλλά με συνοχή πραγματικά, ώστε περίπτωση ιδιαίτερη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των δημοκρατικών αρχών να ενεργοποιήσει αυτή την ε, ύπαρξη παρομοίων όρων και να δούμε και πώς αυτά επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θέλουμε ας πούμε το πάγωμα μιας κάποια συμφωνίας εμπορικής ή όχι από τη στιγμή που έχει κάτι το θετικό σαν αποτέλεσμα και από τη στιγμή που γίνονται σεβαστά αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η προτεραιότητα είναι να δούμε πρώτα απ' όλα πώς, τι αποτέλεσμα έχουν αυτές οι συμφωνίες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα, να δούμε αν είναι κάτι το θετικό ή το αρνητικό. Και από τη στιγμή που θα δούμε αν είναι θετικό ή αρνητικό, να μπορέσουμε σε κάθε περίπτωση χωριστά με συνοχή να συζητήσουμε για τις προϋποθέσεις. Σαν συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέρθηκε ήδη. Αποδείξαμε σε μια έκθεση το καλοκαίρι τώρα ότι η Συμφωνία Επένδυσης και Εμπορίου Ενωμένων Πολιτειών Περού ήταν ε, αρνητικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 33 άτομα βρήκαν το θάνατο και εκατοντάδες άτομα χωρί βρήκαν το, ε, πληγώθηκαν λόγω αυτής της συμφωνίας γιατί έτσι υπήρξαν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των, του ντόπιου πληθυσμού και γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει να δούμε αυτή τη διαπραγμάτευση, τι μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τι μέσα χρησιμοποιήσαμε για να αποδείξουμε ότι η συμφωνία αυτή με το Περού η δική μας ας πούμε δεν θα έχει τα ίδια αποτελέσματα. Είχαμε μια μερική απάντηση γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εμπορική συμφωνία και όχι επένδυσης. Αλλά εδώ και στο μέλλον οι συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε σε κοινοτικό επίπεδο ίσως θα έχουν και την πτυχή επένδυση και χρειάζεται ιδιαίτερα να προσέξουν και θα πρέπει να δούμε την κοινωνική ευθύνη των εταιριών, των επιχειρήσεων, να το προσέξουμε ιδιαίτερα να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αυτό να εκφράσω τη λύπη μου γιατί χρειάστηκε πολύ σύντομα να πάρω το λόγο έτσι πρόχειρα. Είχα προβληθεί κανονικά αργότερα να λάβω το λόγο τη μέρα. Πάντως σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ενδεχόμενα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τερή για όσα μας είπατε και τώρα είναι από την Επιτροπή και πάλι συγγνώμη που αλλάξαμε τη ημερήσια μας διάταξη. Η κυρία Αρνό, μήπως θα ήθελε κάτι να πει σχετικά με τα θέματα που μας απασχολούν. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντρικένε. Θα δώσω με τη σειρά μου ορισμένα στοιχεία που ελπίζω ότι μπορούν να συμβάλλουν τι εργασίε του Κοινοβουλίου. Ε, ε αναμένω όμω ακόμα και άλλου συναδέλφου μου. Απευθυνόμενοι στον κύριο Μάρτιν, νομίζω ότι η συνοχή είναι πράγματι σημαντικό όρο και πρέπει να εφαρμόζεται και πριν από την παρούσα συμφωνία και πριν από τη συνθήκη δηλαδή. Πρέπει να είναι συνεκτική γιατί συχνά έχει ακούσει τη μομφή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρησιμοποιεί διπλά μέτρα και σταθμά. Βέβαια έχουμε διαφορετικά συμφέροντα ανά χώρα. Υπάρχουν βεβαίω ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει και το δικαίωμα βέβαια να αποκτούν ε, οι πολίτες της Ευρώπης ε, πετρέλαιο και φυσικό αέριο και αυτό είναι το ίδιο ε, σημαντικό κατά κάποιο τρόπο έτσι είναι Θε... όπως είπε και ο εκπρόσωπος της ΦΙΝΤΕΑΣ υπάρχει και η θετική αιρεσιμότητα. Ας μην λησμονούμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προσπαθεί να πετυχαίνει την εθελοντική εμπλοκή ε, στις διαδικασίες αυτές των ε, χωρών. Ε, Μία σημαντική έκθεση έκανε πέρσι η κυρία Φλότ σχετικά με τις κυρώσεις. Οι κυρώσεις μπορούν να είναι συμβολικές. Η αποτελεσματικότητά τους αμφισβητείται. Πάντως είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα το οπλοστάσιο μα, οι συνάδελφοί σα και ο κύριο Μάρτιν ιδιαίτερα αναφέρθηκε σε ορισμένα από αυτά. Οι ρήτρε. Εδώ χρειάζεται να κάνω μια μικρή διόρθωση αυτά που είπατε κύριε ε, Μάρτιν. Νομικά οι FTAs, Free Trade Agreements και οι τομεακέ συμφωνίε που μπορεί να είναι αλληλεία ή φορολόγηση κτλ. δεν έχουν πολιτικέ ρήτρε, δεν περιέχουν πολιτικέ ρήτρε όπω η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό που συμβαίνει είναι εκεί όπου έχουμε πολιτικές ρήτρε είναι στο πολιτικό πλαίσιο που είναι για παράδειγμα συμφωνίες εταιρική σχέσης και συνεργασίας. Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα κάπως έχουν περιπλακεί. Ήταν δηλαδή λίγο και εμπόριο, λίγο και κάτι άλλο, λίγο και κάτι άλλο. Ήταν λοιπόν ε, μεικτές συμφωνίες. Όταν έχουμε όμως ξεκάθαρα μία συμφωνία FTA ή sectoral, δεν μπαίνουν ρήτρε. Τώρα αυτό που κάνουμε για να είμαστε συνεκτικοί και όπως ελέγχθηκε από το Κοινοβούλιο και με αρκετή έμφαση, είναι να κάνουμε μία ε, διασύνδεση μεταξύ των δύο. Παράδειγμα Κορέα. Και παράδειγμα οι πρόσφατε συμφωνίε με Περού και Κολομβία. Η FTA έχει μια διασύνδεση με τη Συμφωνία συνεργασία, η οποία περιλαμβάνει τις ε, ε, ουσιώδεις ρήτρες. Πέρυσι είχαμε κάνει ένα σημαντικό εγχείρημα διότι θεωρούσαμε ότι καλά πήγαιναν τα πράγματα ε, ότι, συγγνώμη ότι τα πράγματα πηγαίνανε ε, ε, λίγο από εδώ και από εκεί. Είπαμε στο Κορεπέρ, βάλαμε το Κορεπέρ λοιπόν σε κάθε συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία να μπαίνουν πέντε πολιτικέ ρήτρε και δύο ουσιώδει. Μία από τι ουσιώδει είναι ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δύο λοιπόν ουσιώδει. Γιατί λέγονται ουσιώδει, Διότι συνδέονται με άλλη ρήτρα που είναι η ρήτρα αναστολή. Εάν δηλαδή ε, ε, δεν τηρηθεί η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να ανασταλεί η συμφωνία, η ισχύ τη συμφωνια Αυτή λοιπόν η ρήτρα γίνεται αντικείμενο συστηματικής διαπραγμάτευσης τώρα και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για την ρήτρα, δεν θα έλεγα ότι είναι η πιο πιο πιο σημαντική, αλλά είναι η υψηλότερη γιατί έχουμε πολλές βάσεις στη συνθήκη για την ε, ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όταν ε, διαπραγματευόμαστε τώρα με τις Φιλιππίνες ή με άλλους εταίρους, υπάρχει πολύ μικρό περιθώριο διαπραγματεύσεων ε, για τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι θέλουμε και λέμε και στους εταίρους μας ότι αναφερόμαστε στον χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, των Ηνωμένων Εθνών και στην Παγκοσμία Διακήρυξη Ανθρώπινων Δικαιωμάτων που έχουν συνυπογράψει όλες οι χώρες του κόσμου. Λέμε λοιπόν, κοιτάξτε κύριοι, ποιο είναι το πρόβλημά σας. Εμείς εκεί αναφερόμαστε και βεβαίως συνδέεται αυτομάτως με την ρήτρα αναστολής. Όπως είπε ο συνάδελφος της ΦΙΔΕΑΣ, υπήρξαν 22 περιπτώσεις χρήσης αυτής της ε, πολιτικής ρήτρας αναστολής, 22 περιπτώσεις, αλλά ποτέ δεν υπήρξε πλήρης διακοπή της συμφωνίας. Πάντα ήταν εν μέρη, διότι ό,τι κάνουμε ιδίω για το εμπόριο, πρέπει να είναι και αναλογικό. Μετά λοιπόν από το κούντετα, από το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Αφρική, το είχαμε στο παρελθόν αυτό, αλλά κάθε φορά προσπαθήσαμε να επιτύχουμε ταχύτατο διάλογο. Για παράδειγμα με την Κορέα ήταν ενδεταγμένος ο διάλογος αυτός, διότι φοβόντουσαν οι εταίροι μας ότι θα αποφασίζαμε απότομα να διακόψουμε την ε, εταιρική συμφωνία. Οι χώρε πρέπει να αντιλαμβάνονται ακριβώ περί τίνο πρόκειται. Εμεί του λέμε ότι πολιτικά είναι πολύ σημαντικό, αλλά έχουμε και μια ρήτρα ταχεία ε, συνδιαλλαγής μαζί τους, συνδιαβούλευσης μαζί τους και το άλλο τμήμα της ε, πολιτικής αυτής ρήτρας είναι ότι υπάρχει ε, διάλογος ανθρώπινων δικαιωμάτων. Υπάρχει επομένω θετική εμπλοκή των χωρών. Έχουμε και το ESP που είναι άλλο εργαλείο. Η απόφαση για τη Σρι Λάνκα θα ληφθεί τον Αύγουστο διότι για την ώρα έχουμε μια περίοδο 6 μηνών όπου προσπαθούμε πραγματικά απελπισμένα θα έλεγα να εμπλέξουμε την κυβέρνηση Λάνκα. Όλοι θέλουμε να βελτιωθεί η κατάσταση εκεί. Δεν θέλουμε εν τέλει να αποτύχουμε και εμείς και αυτοί στη βελτίωση της κατάστασης. GSP είναι ένα πράγμα. Εμείς έχουμε διακόψει δύο φορές ήδη την GSP για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Βυρμανία, Μιανμάρ για ε, ε, καταναγκαστικά έργα, λόγω καταναγκαστικών έργων δηλαδή, και με τη Λευκορωσία λόγω ευρύτατης παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τώρα για τη Σρι υπάρχει μια πρόσθετη εμπορική προτίμηση που έχει οδηγήσει σε υπογραφή και κύρωση συνθήκων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το περιβάλλον και για τα δικαιώματα της εργασίας. Προ έγινε μια έρευνα για το Ελσαλβαδόρ. Άρχισε μια έρευνα για το Ελσαλβαδόρ. Πολύ σημαντική άλλωστε, διότι οδήγησε σε αναθεώρηση του, Σαν Σαλβαδοριανού συντάγματος. Άρα, ο στόχος μας δεν ήταν να επιβάλλουμε κάποια τιμωρία στην ε, συγκεκριμένη χώρα, αλλά να καταστήσουμε δυνατό να γίνουν αλλαγέ. Έχουμε λοιπόν και με τη Σρι συνεχιζόμενο διάλογο. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία ή μέσα που διαθέτουμε. Άλλο που συνδυάζεται με το εμπόριο είναι το όμικρον 5 που απαγορεύει το εμπόριο για μηχανήματα, οι ε, ε, συσκευές, ή εργαλεία βασανιστήριων. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Είναι σημαντικό ο κανονισμός αυτός. Δεν είμαι, βέβαιος όμως, δεν βέβαια όμως ε, σήμερα που βρισκόμαστε ε, σχετικά με την εφαρμογή. Επίσης εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού. Γνωρίζετε ότι υπάρχει κοινή θέση υπέρ της ε, μείωσης και της απέτησης εγκρίσεων αδειών για, τον, για το εμπόριο εξοπλισμών σε περιπτώσεις μη σεβασμό ανθρώπινων δικαιωμάτων. Υπάρχει βέβαια και το όπλο των κυρώσεων. Είτε αυτό γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου που θα βασιστεί σε απόφαση του ε, Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και μπορούμε να δούμε αν θα είναι ε, πάγωμα στοιχείων ενεργητικού ή άλλα ε, μέσα ή άλλες κυρώσεις. Όπως είπα Όλοι δεν είναι απαραίτητα ικανοποιημένοι με το ε, όπλο αυτό. Θα αρκεστώ σε αυτά, δεν ξέρω αν ήρθε ο συνάδελφός μου του εμπορίου. Πού είστε. Α, μπορείτε εσείς να συνεχίσετε. Ευχαριστώ. Εγώ θεωρώ ότι η παρουσίαση, η επισκόπηση ήταν πραγματικά εξαντλητική. Δεν μπορώ λοιπόν να προσθέσω πολλά πράγματα. Ακούσατε τα διάφορα όργανα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ακούσατε και παραδείγματα αυτόνομων μέσων, είτε είναι η GSP είτε άλλα. Αποφάσεις που λαμβάνονται μετά από κοινέ θέσεις ε, του Συμβουλίου για διάφορες χώρες. Έχουμε και τα συμβατικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις διμερείς συνθήκες ή συμφωνίες με άλλες χώρες για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την αναστολή της συμφωνίας σε περίπτωση παραβιάσεων κλπ. Και όλα αυτά βασίζονται βέβαια στην ε, πάγια πολιτική διαλόγου με τις ε, διάφορες χώρες. Εγώ προτιμώ να σταματήσω εδώ, εκτός αν έχετε κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα για το εμπόριο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρνό, και ευχαριστούμε και τον συνάδελφό σας. Ερωτήσεις, κύριος Κάζακ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω βουλγαρικά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή η περιβαλλοντική ρήτρα στις εμπορικές συμφωνίες είναι κάτι το πολύ σημαντικό αν λάβει κανείς υπόψη αυτά που μόλις ανέφεραν οι συνάδελφοι. Οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες είναι όλο και περισσότερο είναι όλες και περισσότερες και πρέπει να λαμβάνεται όλο και περισσότερο υπόψη συνεπώς ο αντίκτυπος στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διεθνή ε, συνεργασία για τη δέσμευση των χωρών αυτών στο σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών. Επομένως, ε, πρόκειται για μια πάρα πολύ συνεπή προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερο έχουν κάνει έκκληση για μια τέτοιου είδους συνέπεια καθώς εκλέγονται άμεσα από τους Ευρωπαίους πολίτες. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να παρακολουθούμε τις ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω των ευρωπαϊκών προδιαγραφών που έχουμε θέσει. Άκουσα αυτά τα οποία είπε ο Ντέιβιντ Μάρτιν στην αρχή. Η... Άκουσα τι έχει σκοπό να συμπεριλάβει στην έκθεσή του. Συζητήσαμε τα ζητήματα αυτά και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί να υπάρχουν ε, δύο μέτρα και σταθμά, ότι υπάρχουν ασυνέπειες ε, στην ε, στάση των χωρών ανάλογα με εμπορικά συμφέροντα. Ναι, πράγματι, σε μερικές περιπτώσεις όντως υπάρχει αυτό, σε μερικές φορές, μερικές φορές χρησιμοποιούμε το καρότο και άλλες φορές το μαστίγιο. Πρέπει να ξέρουμε όμως σε τι οδηγεί η μία περίπτωση και σε τι οδηγεί η άλλη. Μετά την έναρξη ισχύω ε, της ε, συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε ότι θέλει να αναλάβει την ευθύνη του ως προς την συνεπή αυτή προσέγγιση. Και έχω ένα ερώτημα να απευθύνω στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε σχέση με τη Σρι Λάνκα και το σύστημα GSP+. Γιατί θελήσατε να το επεκτείνετε στη Σρι Λάνκα και όσον αφορά στην Κολομβία, γνωρίζετε ότι είχαμε μια πολύ εκτεταμένη συζήτηση για την Κολομβία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει σκοπό καν να ξεκινήσει εξεταστική επιτροπή σε σχέση με το κατά πόσο εφαρμόζονται τα κριτήρια. Πολλοί εταίροι, πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, πολλά συνδικάτα έχουν επισημάνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία, όπως επίσης και παραβίαση των κανόνων του ΠΟΕ. Και επομένως θα θέλω να σας ρωτήσω ποιοι είναι οι μηχανισμοί που υπάρχουν. Μιλήσαμε για τους μηχανισμούς ε, επιβολής τέτοιων ρητρών, ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και θα ήθελα να αναφερθώ για παράδειγμα στην συμφωνία με την Κορέα. Μήπως μπορούμε να έχουμε και άλλες νομικές επιλογές, κάποιου είδους μέτρων ε, ασφαλείας εγγυήσεων ώστε να αναστέλλονται οι συμφωνίες αν δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα μπορούσε να είναι υποχρεωτική αυτή η ρήτρα. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Ευχαριστώ πολύ. I will speak in German. Uh, <laughs> θα μιλήσω στα γερμανικά. Τρία πράγματα. Πρώτα, θα υποστηρίξω τον κύριο Μάρτιν για αυτό που λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει έλλειψη συνοχής. Κυρίως όταν, όταν προέρχεται από τη δική μας Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μια εκθέση σχετικά με τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Εξετάστε για παράδειγμα την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία. Εμείς παριστάνουμε σαν δίθεν τα πράγματα να μπορούν να βελτιωθούν από μόνα τους. Μόλις τον Φεβρουάριο ανακαλύφθηκε ε, ο ε, ομαδικός τάφος 2.000 2.000 σωρούς μέσα. Είναι κάτι το απίστευτο. Αυτά τα πράγματα βλάπτουν το κύρος και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Κοινοβουλίου και τη δική μα Επιτροπή, όταν είναι προφανέ ότι χρησιμοποιούνται διπλά μέτρα και σταθμά. Και άλλωστε είναι και εσφαλμένο το μήνυμα που δίνεται στην κυβέρνηση τη Σρι Λάνκα όταν δεν ε, την χάνει ίση μεταχείριση με μια άλλη χώρα. Δεύτερο, η κυρία Νό μίλησε για την έκθεση περί κυρώσεων. Δεν πρόκειται για εμπορική συμφωνία βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό και εν προκειμένου. Δεν ξέρω εάν θα εμφανιστεί στην γνωμοδότηση εάν θα πρέπει να συζητηθεί δηλαδή οι κυρώσει, εφόσον οι κυρώσει αυτέ είναι οικονομικέ κυρώσει, δεν πρέπει να οδηγούν πάλι σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα προσεκτική στο μέλλον θα πρέπει να συζητήσουμε για αυστηρότερε κυρώσει εμπορικές και κατά του Ιράν και μια ερώτηση προ του εκπροσώπους τη Κομισιόν είπατε ότι υφίστανται ιδιαίτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της απαγορεύσεως εξαγωγής εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια. Βέβαια, πολλά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία βασανιστήριων. Αλλά από ό,τι κατάλαβα υπάρχει μια αγορά ηλεκτρικών ε, συσκευών ή εργαλείων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια. Γιατί υπάρχει εκεί ιδιαίτερο πρόβλημα για την παρακολούθηση της ε, αγοράς αυτής και για την εφαρμογή των προβλεπωμένων. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσουν σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θα πω μερικά πράγματα για το GSP, τα, τα, τις ε, βάσεις της σύγκρισης, όπως επίσης και το θέμα της ε, Κολομβίας και της Σρι Λάγκα που ετέθησαν. Το πρώτο που θα έπρεπε να τονίσουμε είναι γεγονός ε, ότι το GSP και τα αυτόνομα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, το θέμα, για τον τομέα αυτό πρέπει να έχουν ε, πολύ αντικειμενικά ε, πολύ αντικειμενική ε, συγκριτική βάση, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύσουν στα πλαίσια διεθνών συμφωνιών και διεθνών κανόνων. Για το λόγο αυτό υπήρχε η επιλογή όταν εγκρίθηκε ο κανονισμός GSP να χρησιμοποιηθεί ε, ε, ένα, να χρησιμοποιηθούν ως βάση διεθνώς αναγνωρισμένες συμβάσεις και νομίζω ότι αυτό είναι η καλύτερη βάση που θα μπορούσαμε να έχουμε. Επίσης έγινε αναφορά σε πολλές ε, συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και συμβάσεων για το περιβάλλον όπως επίσης και για το εμπόριο ανθρώπων. Πρέπει όμως να επεξεργαστούμε περισσότερο την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ε, δράσεων των χωρών ε, που παρακολουθούμε. Αυτή η παρακολούθηση όμως, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει να, έχουμε, πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή να χρησιμοποιούνται τα κριτήρια παρακολούθησης των διεθνών συμβάσεων. Αυτό ε, υπάρχει στον κανονισμό του GSP και επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε πορίσματα του ε, Διεθνούς ε, Οργανισμού Εργασίας, ε, της Αρμοστίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και πολλών άλλων διεθνών οργανισμών. Σε κάθε αξιολόγηση τέτοιου είδους, βέβαια, υπάρχει και ένα πολιτικό κριτήριο και υποθέτω ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το εξαλείψουμε και δεν θα έπρεπε κιόλα, ε, γιατί οι πολιτικοί, οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν την ικανότητα και την ε, εξουσία να λάβουν τέτοιου είδους αποφάσεις και να λάβουν απόφαση βάσει των κριτηρίων που έχουν συμπεριληφθεί στον κανονισμό. Όταν υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα ε, benchmarking που είναι οι συμβάσεις αυτές και υπάρχει παρακολούθηση των διεθνών ε, οργανισμών. Αυτή είναι η βάση επί της οποίας ε, γίνεται, λαμβάνεται η τελική πολιτική απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται με την Κολομβία και τη Σρι Λάνκα τώρα. Δεν πρέπει να μας διαφεύγουν τα εξής ζητήματα. Το GSP Plus είναι ένα πρόγραμμα κινήτρων, δηλαδή δημιουργεί κίνητρα για τις χώρες να βελτιωθούν. Αυτό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην βούληση, την ικανότητα και τη δέσμευση των χωρών ε, στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, ε, αλλά και ε, στη συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση της Σρι Λάνκα, για παράδειγμα, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να διερευνήσει την κατάσταση στη χώρα, δεν υπήρχε συνεργασία και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τι γίνεται με την Κολομβία. Στην... Με την Κολομβία μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων ε, και σοβαρών ε, εσωτερικών συγκρούσεων ε, αποφασίστηκε να τεθούν τα μέτρα και, τα, και οι πολιτικές της Κολομβίας επιτάπητος για εξέταση από τη διεθνή κοινότητα. Δηλαδή η Κολομβία δέχτηκε να παρακολουθείται κάθε χρόνο από, τον, από το σύστημα παρακολούθησης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και είναι τμήμα των καταλόγου των χωρών που τακτικά αξιολογούν σε σχέση με το κατά πόσο τηρούνται οι προϋποθέσεις για την εργασία και για άλλα κριτήρια που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών και επίσης και στο πλαίσιο των οργάνων του ΟΗΕ. Η Κολομβία είπε ότι αυτές είναι ε, αυτή είναι η κατάσταση ε, παρακολουθήστε και δείτε κατά πόσο βελτιώνεται η κατάσταση ή όχι. Σύμφωνα με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βελτιώνεται βέβαια, απέχει πάρα πολύ από το τέλειο, αλλά στο πρόγραμμα των κινήτρων πρέπει να σκεφτεί κανείς ποιες θα είναι οι συνέπειες ε, σε περίπτωση ε, μη εφαρμογής ε, και τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στην συμφωνία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν τα συμπεράσματα των διεθνών οργανισμών, όλοι μπορούν ε, να ε, τα διαβάσουν και να τα κρίνουν. Η άποψη λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι υπάρχουν ε, διεθνή πορίσματα που δείχνουν ότι κινείται η Κολομβία προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι η πολιτική της συνεργασίας με την Κολομβία θα ήταν καλύτερη από τις κυρώσεις και την απομόνωσή της. Θα ήθελα επίσης επί τη ευκαιρία να αναφέρω κάτι που υπόθηκε προηγουμένως σε σχέση με το ε, SIA στο πλαίσιο των ε, διαπραγματεύσεων των εμπορικών και πρέπει να πω ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές βέβαια είναι ανεξάρτητε, γίνονται από συμβούλους, ε, δεν εκφράζουν την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Συμβουλίου των Υπουργών αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους ε, υπεύθυνους διαπραγμάτευσης, όπως επίσης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων. Πρόκειται για αξιολόγηση που εξετάζει τα ζητήματα της απελευθέρωσης του εμπορίου και των δεσμεύσεων για το εμπόριο σε βασικούς τομείς, όπως είναι η μείωση της φτώχειας, η πρόσβαση σε ε, υγειονομική ε, υγειονομική υποδομή όπως επίσης και για ζητήματα δημόσιας υγείας, κοινωνικά δικαιώματα, ε, θέματα που έχουν να κάνουν ε, σε μεγάλο βαθμό με ε, οικονομικά ζητήματα, μεταρρύθμιση πολλών τομέων, κάτι που να δείχνει το άνοιγμα της χώρας. Η Πρόεδρος διακόπτη, μήπως μπορείτε να συνοψίσετε. Ναι, αυτό θα έλεγα, δεν ξέρω αν για τα βασανιστήρια θα ήθελε η κυρία Αρνό να προσθέσει κάτι. Ακούστε για τα βασανιστήρια. Μια επιτροπή τακτικά συνεδριάζει για να δει την εφαρμογή του εργαλείου αυτού και όπου το θέμα είναι ότι ο κατάλογος αυτών των θεμάτων που υπάρχει σε αυτόν τον κανονισμό και το σκεφτόμαστε πώς θα πρέπει να διευρύνουμε αυτόν τον κατάλογο και είναι αρκετά περίπλοκο πάντως. Κάτι που ήθελα να πω σχετικά με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν παίρνουμε μια χώρα και λέμε είναι στο αυτό το επίπεδο ή στο ίδιο επίπεδο. Ε, κοιτάμε το εμπόριο. Κοιτάζουμε και την τάση μετά και με την Κολομβία. Αυτά που είπατε είναι σωστά. Έχουμε πολλούς ε, πολλές εισηγήσεις από τα δεδομένα Έθνη και σε διεθνή βάση και οι εισηγητές είπαν αυτό, αυτό και αυτό συμβαίνει και νομίζομαι ότι προχωρούν εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε και αυτά που είπε ο κύριος Μάρτιν ότι τώρα πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια μελέτη και ήρθε στο τέλος του χρόνου στο Κοινοβούλιο για το εμπόριο και τις διάφορες ελευθερίες. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο τίθεται πάντα, το θέμα του εμπορίου με ε, ε, προϊόντα τα οποία παράγονται στη φυλακή. Εδώ ακριβώς για όλη τη σκέψη, για όλο το συλλογισμό με το Κοινοβούλιο σχετικά με την έκθεση αυτή που ο κύριος Μάρτιν ε, συντάσσει θα πρέπει να δούμε και τη μεταφορά τεχνολογίας που ξέρετε ότι με τα θέματα ας πούμε της Κίνας και το πώς ορισμένοι είχαν τη δυνατότητα μια κάποια στιγμή να κάνουν ένα έλεγχο στην πρόσβαση στο ίντερνετ νομίζω ότι θα θα όλο και περισσότερο αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει μια λύση και έχουμε συνειδητοποιήσει βέβαια ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που θα πρέπει να ελέγξουμε. Το θέμα δε της συνοχής ε, μας απασχολεί. Σας ευχαριστώ. Thank you. Thank you, Ευχαριστούμε. Κύριε Μάρτιν. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους μου και την Κομισιόν και τον κύριο Τερή για τα χρήσιμα που μας είπαν. Ο κύριος Τερή είπε σχετικά με την μελέτη επιπτώσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ νομίζω ότι είναι σωστό. Θα πρέπει να γίνει μαζί με την μελέτη επιπτώσεων, οικονομικών επιπτώσεων δηλαδή που κάνουμε για όλες τις FTA και δεν ξέρω αν ενθουσιάζει κάτι τέτοιο τις χώρες μέλη, αλλά ως κοινοβούλιο μπορούμε να το κάνουμε αυτό ανάμεσα στην μονογραφή της συμφωνίας και στην ε, χορήγηση εγκρίσεως του Κοινοβουλίου. Να δούμε δηλαδή εάν ένα, ε, μια συμφωνία FTA είναι ε, καλή ή κακή πρόπτικη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συζήτηση Σρι Λάνκα κατά Κολομβίας ήταν χρήσιμη. Θα δούμε τώρα. Υπάρχει πάντως κοινό έδαφος μεταξύ Κομισιόν και μου και του Κοινοβουλίου ότι βέβαια τα benchmarks της GSP πρέπει να είναι βασισμένα σε διεθνείς ε, συμφωνίες, σε διεθνεί συνθήκες. Ασφαλώς και πρέπει ε, να ε, γίνεται monitoring και από αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς. Πώς ερμηνεύονται όμως αυτές οι διεθνείς συμφωνίες και πού αρχίζουμε να διεξάγουμε έρευνα ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα εμείς και ποια στιγμή παραμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα επαναλάβω αυτό που είπα και πριν και που επιβεβαιώθηκε από τον δεύτερο εκπρόσωπο της Κομισιόν ότι είναι περισσότερο μια αίσθηση της ε, Κομισιόν για το προς τα που πηγαίνει μια χώρα. Η Σρι δεν ε, ήθελε να μπει σε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Κολομβιανοί ναι, είναι όμως γνήσιος ο διάλογος ή μήπως είναι επιφανειακός. Μήπως απλώς έχουν καλύτερες δημόσιες σχέσεις οι Κολομβιανοί από τους Σρι Μπορεί και να μην είναι έτσι βέβαια και ελπίζω να μην είναι έτσι. Αυτό που νομίζω πάντως ότι δείχνουν όλη, όλα τα σχετικά στοιχεία είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει ως διεθνής κοινότητα, ως ευρωπαϊκή κοινότητα μάλλον, να εξετάσουμε την κατάσταση στην Κολομβία και μετά να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μερικά τα στοιχεία, είναι ε, ε, ε, εν μέρη μόνο ασφαλής οι εκτιμήσεις μας. Και πάλι κάπου όπου φάνηκε να συμφωνούμε είναι ότι χρειάζεται περισσότερη συνεκτικότητα και συνοχή. Τι είναι συνεκτικό και τι είναι συνεπές. Θα μου πει βέβαια η πρόεδρος να ολοκληρώνω. Ναι, η πρώτη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε και για τις άλλες συμφωνίες, για τα βασανιστήρια κτλ. Αυτά θα πρέπει να μπουν και στη γνωμοδότησή μας. Και, υπάρχουν και υπάρχει και ένα έγγραφο του που αυτή τη στιγμή συντάσσεται στην ε, Επιτροπή Εμπορίου και αν μπορέσουμε να το βάλουμε μέσα, τόσο το καλύτερο. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Όσοι ενδιαφέρεστε, να γνωρίζετε ότι θα συζητήσουμε την εφαρμογή των κανονισμών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Μαρτίου σε ό,τι αφορά δηλαδή την απαγόρευση εξαγωγής ε, εργαλείων ε, ή συσκευών που χρησιμοποιούνται σε βασανιστήρια και υπενθυμίζω στους συναδελφούς το χρονοδιάγραμμα που έχει ως εξή. συζήτηση του σχεδίου γνωμοδότησης στην Υποεπιτροπή προβλέπεται για τις 26 και 27 Απριλίου Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 28 Απριλίου στις 6 το απόγευμα. Συζήτηση τροπολογιών στην Υποεπιτροπή 10 Μαΐου. Ψήφος στην Επιτροπή Εξωτερικών στις 31 Μαΐου έως 2 Ιουνίου. Επίσης η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Απασχόλησης και Ανάπτυξης, αυτές οι επιτροπές πρόκειται επίσης να καταθέσουν γνωμοδοτήσεις. Ευχαριστώ όλες και όλους όσοι έλαβαν το λόγο. Θα προχωρήσουμε στην ακρόασή μας τώρα για την άσκηση βίας κατά γυναικών σε περιπτώσεις ενόπλων συγκρούσεων. Έχουν προσέλθει πολλά πρόσωπα για να συμμετάσχουν στην ακρόαση αυτή. Καλώς ήρθατε όλες και όλοι. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων εντάσσεται στο πρόγραμμα του εορτασμού της α, ημέρας της γυναίκας, της Εθνούς ημέρας της γυναίκας, στις 8 Μαρτίου. Οι προσκεκλημένοι μας έχουν συμμετάσχει και σε άλλες εκδηλώσεις την εβδομάδα αυτή. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να επισκεφθείτε στον τρίτο όροφο φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Ο βιασμός ως ο πολεμικό όπλο στην περίπτωση των γυναικών του Κονγκό. Στους ομιλητές μας έχουμε πει ότι θα έχουν για τις παρεμβάσεις τους περίπου 10 λεπτά. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να μην υπερβείτε το όριο αυτό. Η κυρία Χάουζερ και η κυρία Ζιμπαμπού έχουν εμπειρία σχετικά με την παροχή φροντίδων σε γυναίκες που έχουν υποστεί ε, ψυχολογικούς και άλλους τραυματισμούς από τέτοιες ε, ε, περιπτώσεις και υπάρχουν και άλλα πρόσωπα εδώ που έχουν ανασχοληθεί με την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του, των Ηνωμένων Εθνών καθώς και με άλλα θέματα κατευθύνων γραμμών για την αντιμετώπιση της βίας κατά γυναικών. για την εφαρμογή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση του ψηφίσματο τη Γενική Συνέλευση ε, ε, των Ηνωμένων Εθνών για τα ψηφίσματα 1325 και 1802 και ναι μεν οι κατευθυντήριες γραμμές ε, και το φάσμα εφαρμογής τους υπερβαίνει την βία κατά γυναικών σε πολεμικές συγκρούσεις αλλά και περιλαμβάνει και την βία ε, κατά γυναικών οίκη, δηλαδή ε, στις αιστείες τους ε, θα δούμε τι θα μας πούν η κυρία Χάουζερ πρώτα ιδρύτρια και επικεφαλής της, Μοντικα, της Μοντιάλ έχετε το λόγο Μάλιστα θα σας ευχαριστήσω πρώτα στη γερμανική γλώσσα για την πρόσκληση που απευθύνατε σε μένα και στη συναδελφό μου Ζανίν Μουκανέβα για να μιλήσουμε για ε, περιπτώσεις γυναικών που έζησαν και επέζησαν στο παράδειγμα εδώ του Ανατολικού Κονγκό ε, σεξουαλικές επιθέσεις και ελπίζω να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό όχι βέβαια μόνο με την αφορμή της 8ης Μαρτίου μαζί με Βόσνιες συναδέλφους ίδρυσα προ 17 ετών την οργάνωση Medica Mondial. Δεκάδες χιλιάδες γυναικών έπεσαν τότε θύματα βιασμών. Φτιάξαμε λοιπόν μια οργάνωση που θεωρούσαμε ότι έλειπε για την παροχή υποστήριξη και ανθρωπιστική βοήθεια σε γυναίκες οι οποίες έχουν ζήσει τέτοιες εμπειρίες. Σε αυτά τα 17 χρόνια ε, έχουμε κάνει advocacy, έχουμε, κάνει, έχουμε αναπτύξει αρχές και ε, τρόπους αντιμετώπισης των ψυχολογικών τραυματισμών. Συνεργαζόμαστε από το 1996 και με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης και διερωτώμεθα συνεχώς τι σημαίνει για τις γυναίκες η δικαιοσύνη. Από πολλά χρόνια ε, συμμετέχουμε σε σχέδια στα Βαλκάνια, επίσης από το 2002 στο Αφγανιστάν, επίσης στην Λιβερία και σε άλλες ε, περιπτώσεις κρίσεων και στην Γκόμα με την ε, οργάνωση ΠΑΙΦ. Για μένα είναι πραγματικά επώδυνο και ανυπόφορο παρόλο τα ψηφίσματα να μην έχουν βελτιωθεί, να μην έχει βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών σε ε, παιδεία συγκρούσεων. Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Συγκρούσεις στο Ανατολικό Κογκό κάνουν ε, άνδρες οι οποίοι διψούν για εξουσία και χρησιμοποιούν την ε, βία αλλά και τους βιασμούς κατά γυναικών και κοριτσιών για να καταστρέψουν τις ίδιες τις οικογένειές τους και τις κοινωνίες τους και αυτό τραυματίζει τις γυναίκες για το υπόλοιπο της ζωής τους, ενώ οι δράστες σπάνια, σπανιότατα διώκονται. Αντιθέτως με τον πόλεμο της Βοσνίας, σήμερα έχουμε το ψήφισμα 1325 των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο θεσπίζει ίσα δικαιώματα των γυναικείων πληθυσμών για ε, συμμετοχή τους σε, ειρηνικές, σε ειρήνης. Και από το ε, ψήφισμα 1820 μόλις έχουν περάσει λίγα χρόνια το οποίο είχε ως στόχο να ε, προστατευτούν οι γυναίκες απέναντι στους βιασμούς. Υπάρχει και διεθνές δικαστήριο το οποίο έχει δημιουργηθεί για να επιβάλλει ποινές στους δράστες τέτοιων εγκλημάτων και να πάψει η ατιμορρησία. Όμως, σύμφωνα με το Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών παραπάνω από 100.000 γυναίκες και κορίτσια ε, βιάστηκαν με τον πιο βάρβαρο τρόπο το 2008. Πάνω από 20% των γυναικών δε μολύνθηκαν με τον ιό του AIDS. Όλοι συμμετέχουμε στην προσπάθεια αντιμετώπισης. Για όλους και όλους είναι σημαντικό να αλλάξει η κατάσταση γυναικών στις περιπτώσεις κρίσεων. Ο ίδιος ο Κογκολέζικος στρατός και η Εθνική Αστυνομία ευθύνονται. Η τόπια στρατηγική των ομάδων αυτών υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκεται όμως σε λάθος βάση η ανάλυση των δεδομένων. Ο βιασμός σε βάρος γυναικών και κοριτσιών αντιμετωπίστηκε για πολλά χρόνια σαν αποκλειστικό πρόβλημα των γυναικών, όπως στην πραγματικότητα είναι πρόβλημα ανδρικό και είναι πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Παρόλο το έργο πολλών εμπνευσμένων Κογκολέζων και στο εθνικό και στο διεθνές επίπεδο το πρόβλημα των βιασμών παραμένει σοβαρό και μέσα στα πλαίσια της ειρηνευτικής διαδικασίας. Υπήρξαν βέβαια κάποιες φωνές που ακούστηκαν κατά της ατιμορρησίας αλλά δεν έχει γίνει αποτελεσματική προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Η εντολή της ΜΟΝΙΟΚ, της Δύναμης των Ηνωμένων έχει κατά προτεραιότητα την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Ωστόσο, δεν βρίσκεται στην πραγματικότητα στο ε, πυρήνα των προσπαθειών της μονούκ Η κατάσταση είναι παράξενη και δείχνει πόσο είναι απελπισμένες οι προσπάθειες ε, των οργανώσεων γυναικών για να προστατεύσουν τις κογκολέζες γυναίκες και κορίτσια τοπικές οργανώσεις γυναικών προσπαθούν να πιέζουν μάλλον για να θεσπιστεί εθνικός νόμος στο Κονγκό για να προστατεύονται οι γυναίκες και τα δικαιώματά τους. Ακόμα, ωστόσο, δεν υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη μέσα στα πλαίσια της ΜΟΝΟΚ που να συλλαμβάνει και να άγει ενώπιον της εθνικής δικαιοσύνης τους δράστες. Το παράδειγμα της Λιβερίας είναι εντυπωσιακό. 600 γυναίκες αστυνομικοί από την Ινδία υποστηρίζουν τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ, συλλαμβάνουν τους δράστες και τους άγουν ενώπιον της εθνικής δικαιοσύνης, συλλέγουν δέντα σχετικά στοιχεία για ε, να γίνει η δίωξη. Ένα θαυμάσιο παράδειγμα το οποίο μπορεί να ε, γίνει και μέσα στα πλαίσια της ΜΟΝΟΚ η Μονούκ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύσουν τις γυναίκες απέναντι στους βιασμούς. Η νέα εντολή της Μονούκ πρέπει να περιλάβει ρητά την προστασία κατά των βιασμών και όλα τα rules of engagement πρέπει να περιλαμβάνουν το ίδιο. Αυτό που θα σημάνει στην περίπτωση αυτή είναι το εκόλουθο παράδειγμα από την Γκόμα. Οι εταίροι μας της ΠΑΙΦ προσπάθησαν ξανά και ξανά να επιτύχουν την υποστήριξη της Μονούκ αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών για να απελευθερώσουν κορίτσια τα οποία είχαν εχμαλωτιστεί για να ε, χρησιμοποιηθούν ως ε, στην πραγματικότητα για την γενετήσια ικανοποίηση των μελών των πολιτοφυλακών. Πήγαν να διαπραγματευτούν με επικίνδυνους επικεφαλείς των πολιτοφυλακών για να απελευθερώσουν τα κορίτσια. Κάθε φορά που το κάνουν αυτό, οι ίδιες αυτές οι εκπρόσωποι κινδυνεύουν να βιαστούν και να φωνευτούν. Σας ρωτώ λοιπόν, γιατί έχουμε κατευθύνες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστατεύονται οι διάφορες ακτιβίστριες εάν δεν εφαρμόζονται. η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει για την εφαρμογή των οδηγιών της δυνάμεις προσωπικό για να παρακολουθεί τις δίκες, να εγγυάται δίκες δίκες και να δώσει ένα καθαρό μήνυμα στην κυβέρνηση του Κονγκό ότι πρέπει να σέβεται τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Θα πρέπει να πιεστεί η κυβέρνηση του Κονγκό να σέβεται τους εκπροσώπους ε, οργανώσεων ανθρωπινών δικαιωμάτων που συχνά κρατούνται αυθαίρετα και αντιμετωπίζουν απειλές και ιδίω όταν θα συζητηθεί ξανά η εντολή των δυνάμεων της Μουνιούκ. Για το λόγο αυτό, για το σκοπό αυτό, ζητούμε να υποστηριχθεί η κοινωνία των πολιτών στις συζητήσεις αυτές. Δεύτερο, η προστασία κατά του βιασμού και άλλων μορφών βίας κατά των γυναικών να αποτελέσει μέρος των διμερών και πολυμερών συμφωνιών σχετικά με μια στρατηγική εξόδου με τον ε, πρόεδρο Καμπίλα και τους αξιωματούχους του. Επίσης, οι οργανώσεις βάσης των γυναικών να επωφελούνται περισσότερο από τα χρήματα που προσφέρουν οι δωρητές. Τα χρήματα αυτά πηγαίνουν κυρίως στις μεγάλες ανθρωπιστικές οργανώσεις. Οι μικρές μη κρατικέ οργανώσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν μεγάλα ποσά από του προπολογισμού αυτού. Το Ευρωπαϊκό Μέσο Δημοκρατίας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων είναι σημαντικό όργανο για πολλές περιοχές και χώρες που βρίσκονται σε κρίση. Θα ήθελα να πω όμως ότι για τις μικρές οργανώσεις βάσης υφίστανται πολλά τεχνικά προβλήματα για να υποβάλουν αιτήσει για να απολαύσουν ποσά από τα χρήματα αυτά. Όμως αυτές οι μικρές οργανώσεις είναι σημαντικές γιατί υποστηρίζουν θύματα βιασμών επιτόπου και ταυτόχρονα είναι οι οργανώσεις εκείνε οι οποίες καλούνται να εργαστούν και να λειτουργήσουν υπό την διαρκή απειλή των κυβερνητικών εκπροσώπων των περιοχών αυτών και των πολιτοφυλακών. Πρέπει να μπει ένα τέλο επιτέλου στους βιασμού και στη συνάσκηση βία κατά γυναικών. Η ατιμορρησία είναι ένας από τους μεγαλύτερους λόγους ανησυχίας στην λαοκρατική δημοκρατία του Κονγκό. Μπορούν να εφαρμοστούν όμως και εκεί παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτιάξει ένα νοδικό χάρτη για τη βελτίωση και για την ε, αναδιάθρωση της δικαιοσύνης. και να μπουν στον πυρήνα των πολιτικών αυτών τα μέτρα για την προστασία των γυναικών να γίνεται διαβούλευση με τις οργανώσεις των γυναικών ώστε η εφαρμογή να είναι αποτελεσματική. Τέλος, δίδω ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι το πρόβλημα των βιασμών σε περιπτώσεις συγκρούσεων είναι ενδυμικό και σε μεγάλη κλίμακα, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι χρειάζεται μια εκπρόσωπο η οποία να ασχολείται ειδικά με το θέμα αυτό, για να υπάρξει και μεγαλύτερο αποτέλεσμα συνέργειας με τις διάφορες άλλες ε, μονάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες καλούνται σε όλες τις εκπροσωπήσεις των γυναικών να γίνουν προσπάθειες για να προστατεύσουν τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια από την άσκηση βίας σε βάρος τους. Αν θέλουμε πραγματικά να σταματήσουμε τα εγκλήματα αυτά, χρειαζόμαστε την τεχνογνωσία που έχουν οι οργανισμοί αυτοί. Να δούμε επίσης πώς θα γίνει διασύνδεση και με άλλα προγράμματα όπως προγράμματα ασφάλειας, βελτίωση της διακυβέρνησης και ούτω καθεξής. Το 2009 καταδικάστηκαν 10 βιαστές στην κόμμα από ε, κογκολέζικο στρατοδικείο. Πώς κατέστη αυτό δυνατόν. Για τους εξής τρεις λόγους. Διεθνής δράση των Ηνωμένων Εθνών μετά την επίσκεψη της Χίλαρη Κλίντον στην Κινσάσα, όπου τους τα είπε πάρα πολύ ξεκάθαρα. Δεύτερον, συνεχής awareness raising από ντόπιε μη κρατικέ οργανώσεις και τέλος με τις προσπάθειες και τις μαρτυρίες των γυναικών εκείνων που επέζησαν αυτών των ε, ε, βιασμών οι οποίες μπόρεσαν έτσι να συμβάλλουν στην απονομή της δικαιοσύνης. Αφού αυτές οι κοπέλες και αυτά τα κορίτσια μπόρεσαν να μιλήσουν παρά τον φόβο εκδίκησης παρά τον καθημερινό, το καθημερινό στίγμα που θα φέρουν, τότε εμείς πρέπει να τις ενισχύσουμε και να συμβάλλουμε στην απονομή δικαιοσύνης για την αξιοπρέπεια και των θυμάτων και τη δική μας αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάουζερ για όσα μας είπατε. θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε και σε ερωτήσεις. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω την ομιλήτριά μας από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ζανίν Τσιμπάμπου Μουκανίγουα, ε, συντονίστρια του προγράμματος ΠΑΙΦ. Έχετε το λόγο. Euh, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα συμπληρώσω την προηγούμενη ομιλητή, την προηγούμενη ομιλήτρια. Εδώ η κατάσταση για τη γυναίκα στις χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση είναι ίδια σε όλες τις χώρες. Κυρίως βιασμό, ε, σεξουαλική ομοιρία, και αυτά σε όλες τις χώρες, στις χώρες του Βορρά αλλά και του Νότου ταυτόχρονα, εκεί που έχουμε ένα πόλεμο, από αυτά τα δεινά υποφέρουν οι γυναίκες. Θα σας πω στο δικό μου κράτος τι ακριβώς συμβαίνει για τη γυναίκα. Λοιπόν, Εμεί βγήκαμε από τον πόλεμο, ξεφύγαμε από τον πόλεμο και υπάρχει μια διαφάνεια δημοκρατική και έτσι έχουμε τα θεσμικά όργανα, ε, τα δημοκρατικά και οι γυναίκες ε, και γύρω τους διεξάγεται ακόμα ένας πόλεμος, συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Είναι ο ίδιος ο στόχος των ένοπλων ε, ομάδων ε, σε ανταγωνιστικό επίπεδο που είναι στις ανατολικές επαρχίες ε, και στις βορειές επαρχίες. Α, λοιπόν, σεξουαλική βία που χρησιμοποιείται σαν στρατηγική πολεμική για να καταστρέψουν οι οικογένειες στην τοπική κοινωνία και το σύνολο του έθνους μας. Οι γυναίκες ήδη υποφέρουν και ακόμα μια φορά βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουν ένα φαινόμενο σεξουαλικού εγκλήματος παρά το ότι έχουν υιοθετηθεί πάμπολα ψηφίσματα από το Σύμβουλο Ασφαλείας των Εθνών. Το 13-25 ψήφισμα, 10 χρόνια ήδη, το 18-20 ψήφισμα, 2 χρόνια, αλλά παραμένουν ατιμόρυτα τα εγκλήματα αυτά. Παρά τις προσπάθειες ε, της κυβέρνησης του Κονγκό σε νομικό επίπεδο, της έγκρισης ε, του νόμου για την καταστολή του σεξουαλικού εγκρήματος ε, και της διάκρισης λόγω του φύλου, παρόλα αυτά εξακολουθούν ε, να υπάρχουν ε, αυτά τα εγκλήματα κατά των γυναικών. Η απάντηση της διεθνούς κοινότητας μέσω των ε, οργάνων του ΟΗΕ, της UNIFEM, των μη κυβερνητικών οργανώσεων των διεθνών, αλλά και των τοπικών φορέων, ήταν ότι πρόκειται για ζητήματα επίγοντα Επίσης ε, υπάρχουν και πολλές προκλήσεις ε, γιατί τα θύματα της κατάστασης αυτής ε, είναι δύο φορές θύματα, επιτρέψτε μου να πω. Δεν είναι μόνο θύματα ε, λόγω αυτού που υφίστανται, αλλά επίσης στιγματίζονται και στην τοπική κοινότητα. Τα κονδύλια για την καταπολέμηση της μάστιγας αυτής δεν φτάνουν στα θύματα. Γιατί τα θύματα ζουν σε, ε, στην Ήπεθρο όπου δεν υπάρχουν ε, ε, υγειονομικές εγκαταστάσεις για να τις βοηθήσουν ε, και δεν υπάρχουν επίσης και... δεν υπάρχει και δικαιοδοσία για την εκδίκαση των εγκλημάτων αυτών. Και όπως σας είπα και προηγουμένως υπάρχει μια πρόκληση, πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε προκειμένου να αναλάβουμε, προκειμένου να ε, αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα αυτή. Μέχρι τώρα περισσότερο τις συνέπειες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και όχι την αιτία που είναι κυρίως η ασφάλεια, η έλλειψη ασφάλειας στο ανατολικό τμήμα της χώρας αν υπάρχουν προγράμματα και προσπάθειες που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει την ε, γυναίκα στο Κονγκό, ε, αυτό αφορά πραγματικά τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασφαλείας, όπως κάναμε και με τη μεταρρύθμιση του ε, νομικού συστήματος. Βέβαια παραμένουν πολλά που μπορούν να γίνουν ακόμη. Υπάρχουν ακόμη επαρχίες στις οποίες Έχουμε καταδικάσει πολλούς, ε, αλλά δεν υπάρχουν φυλακές να, τις βάλουμε, να, τους, ε, να τους βάλουμε μέσα. Δηλαδή κυκλοφορούν ελεύθεροι, έχουν μεν καταδικαστεί ως εγκληματίες, αλλά ε, δεν είναι σε, θέση οι φυλακές να στεγάσουν όλους αυτούς ε, τους ανθρώπους. Η ατιμορρησία όμως συνεχίζεται. Σήμερα, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, από το 2002 επιλαμβάνεται τέτοιων ζητημάτων, όμω, τόσα χρόνια είναι σε ε, πόλεμη κατάσταση η χώρα και εξακολουθούν τα ζητήματα αυτά να μην αντιμετωπίζονται. Πότε επιτέλους το θέμα της, ατι... θα αντιμετωπιστεί και πότε θα σταματήσουμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί οι υπεύθυνοι, οι δεράστες ε, των εγκλημάτων ε, αυτών ε, από το 1976 μέχρι το 2002 δεν θα τιμωρηθούν και αυτό είναι απαράδεκτο για τις γυναίκες του Κονγκό. Επίσης υπάρχει και το θέμα της αποκατάστασης των θυμάτων. Γιατί είναι κάτι που τις πλήττει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ε, παραβιάζεται το σώμα τους, ε, ακροτηριάζεται, ακροτηριάζονται τα, τα γενετικά τους όργανα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταματήσει. Υπάρχει και αυτή η πτυχή που είναι πολύ ευαίσθητη και πρέπει να ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα διάφορα προγράμματα ε, στο, που... αναλαμβάνει για τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Υπάρχουν ε, οι τοπικές ε, και οι ξένες ε, δυνάμεις και οι γυναίκες αποκλείονται. Αν δούμε το ψήφισμα 1325, οι γυναίκες κανονικά θα έπρεπε να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίλυση των διαφορών και ότι πρέπει να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις ε, στο πλαίσιο της χώρας. Και μάλιστα υπήρξαν και σχετικά όργανα που δημιουργήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Η παρουσία των γυναικών πολλές φορές αλλάζει ακόμη και τη φύση των συμφωνιών. Και πρέπει πάρα πολύ να δουλέψουμε για τα ζητήματα αυτά, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να συμμετέχουν στην ε, εδραίωση της ειρήνης, γιατί σε αυτή ακριβώς την φάση βρίσκεται η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Ένα πρόβλημα, μία ακόμη πρόκληση είναι οι πρωτοβουλίες ε, ειρήνης ε, των γυναικών ε, σε χώρες που βρίσκονται σε ένοπλες συγκρούσεις. Μιλάω για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, όπου βρίσκεται και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν επιδοτήσεις για τις γυναικείες πρωτοβουλίες, γιατί ο προϋπολογισμός, τα προγράμματα ε, των γυναικών ε, στις ε, χώρες αυτές δεν χρηματοδοτούνται. Η χώρα των μεγάλων λιμνών, το Μπουρούντι, η περιοχή των μεγάλων λιμνών, το Μπουρούντι, η Ρουάντα και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ήδη τέτοιου είδους προγράμματα, ε, όπως προβλέπει το ψήφισμα 1325 αλλά για να ε, εφαρμοστούν τα προγράμματα αυτά πρέπει να υπάρξει κάποια στήριξη. Χρειάζεται οικονομική στήριξη. Και γι' αυτό ακριβώς ε, έτσι θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου με την έκκληση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Μπεατρίς Λορέντζο είναι η επόμενη ομιλήτρια μας ε, από την Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, που εκπροσωπεί την Ισπανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Από την Ισπανική Προεδρία είναι τιμή για μένα να παρεμβρίσκομαι εδώ για, να... για τις συζητήσεις αυτές και για τις κατευθυντήρες γραμμές ε, για την ε, διακάλυψη των γυναικών και τις διακρίσεις εναντίον τους ε, για τα ισότητα μεταξύ των δύο φύλων από οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής πλευράς. Ε, έχουμε εκεί ένα πυλώνα κεντρικό της κυβέρνησής μου αυτά τα τελευταία χρόνια και δείχνει ακριβώς με τον άξονα ε, που έχει να κάνει με όλη τη δράση εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φάνηκε καθαρά με την έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το θέμα αυτό και με διάφορα εσωτερικά μέτρα που έχουν ληφθεί ενάντια στην βία κατά των γυναικών. Στην εξωτερική δράση δε έχουμε προστασία των γυναικών στα πλαίσια έμεσα σε κάθε μία από τις οκτώ κατευθυντές γραμμές Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την κατάσταση που επικρατεί στις γυναίκες που ε, βρίσκονται σε κίνδυνο σε κάθε μέρος του κόσμου και η βία κατά των γυναικών και των μικρών κοριτσιών με τη διάκριση που υπάρχει εναντίον τους είναι το πιο διαδεδομένο έγκλημα στον κόσμο όπως ακριβώς φάνηκε καθαρά στις συζητήσεις εδώ. Και εδώ το Δεκέμβριο του 2008 είχαμε μια κατευθυντήρια γραμμή που υφετήθηκε που αποκλειστικά ε, μάχεται κατά του προβλήματος αυτού σε μια ευρεία έννοια ακριβώ ε, της μάχης αυτής ε, που αναφέρεται σε οποιαδήποτε είδος βίας το οποίο απορρέει και καταλήγει σε σεξουαλικές ψυχολογικές ζημιές στη γυναίκα όπως επίσης και απειλές για πραγματοποίηση παραγωγικών πράξεων. Είναι μια έννοια που προχωράει πολύ περισσότερα από την άχηση βίας κατά των γυναικών στα πλαίσια, των, ε, στα πλαίσια εχθροπραξιών και εμπολεμής κατάστασης. Η Ισπανία είναι το τρίτο κράτος που ε, προσπαθεί να εφαρμόσει αυτές ε, τις κατευθυντικές μετά από τη Σουηδική και την Τσεχική Προεδρία. Εδώ έχουμε ολοκληρώσει μια πρώτη φάση αυτής της κατευθυντικής γραμμής και η κατευθυντήρια αυτή γραμμή αρχική βοήθησε και μάλιστα τώρα τα τελευταία δύο έτη πέρα από ότι εφαρμόστηκε άμεσα και τάχιστα πρώτα απ' όλα ενημερώσαμε τις πρεσβείες, τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ε, και την κοινωνία των πολιτών για την εφαρμογή όλων αυτών, όπως επίσης και ένα διάλογο ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και στις πρεσβείες, το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι κατευθύνες γραμμές και επίσης ε, πληροφορίες ε, γενικά για την συγκεκριμένη κατάσταση επιτόπου για να λάβουμε και από πλευράς πρεσβειών και αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε εκθέσεις για 88 χώρες και στα πλαίσια αυτής της άτυπης ομάδας ε, η ΚΟΧΟΜ η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Task Force που ασχολείται με αυτά ανέλησαν ε, αυτές τις 88 εκθέσεις μαζί με τις πληροφορίες που περιέχονται και αυτά, σε αυτά σε ένα ευρύ κατάλογο, τον κύριο κατάλογο όπως αποκαλείται και ο οποίος εφαρμόζεται και εξετάζεται και ακριβώς ε, Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία πολύτιμα για τη δουλειά σε αυτό το τομέα και είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης και των πρεσβειών επιτόπου και για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται από τις κατευθυντήρες γραμμές. Πάνω σε αυτά ακριβώ η Ισπανία, έχοντα την Προεδρία αυτό εξάμεινο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προώθησε, θα προωθήσει πάντα τα εξή μέτρα. Καταρχήν, αυτός ο πίνακας να είναι ένα βασικό κείμενο που θα ενημερώνεται, θα συμπληρώνεται από τις πρεσβείες και από την κοινωνία των πολιτών επιτόπου και ο στόχος θα είναι στην ενημέρωση αυτή, στην πληροφόρηση αυτή να είναι η πραγματικότητα και να μπορέσει να διευκολουθούν οι ενέργειές μας. Ακόμα προχωράει η σύσταση ε, σχετικά με την ε, με τις πληροφορίες αυτές σε περιφερειακό, γενικό, εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο ήδη δώσαμε οδηγίε της πρεσβείας μας να εφαρμόσουν αυτές τις συστάσεις, τις συγκεκριμένε που έχουν συμπεριλάβει στις εκθέσεις τους και που από τις ομάδες εργασία μας υιοθετήθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο αυτές, ε, αυτός ο πίνακας ε, και Αυτές οι εκθέσεις θα πρέπει να θετηθούν για συστάσεις επίσης περιφερειακού χαρακτήρα που να μπορούν να εφαρμόζονται σε διάφορες περιοχές του κόσμου και ταυτόχρονα θα έχουμε διάφορες γενικές συστάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εφαρμοστούν σε πλευρές επαφές και επίσης εφαρμογή στρατηγικών περιφερειακών από πλευρά πρεσβειών μα ε, και επιτόπου, εκεί που θεωρούν ότι είναι απαραίτητο και σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Επίση, προθεσμία δύο ετών μέχρι το 2012 για την επεξεργασία αυτών των στρατηγικών και μετά οι πρεσβείε και οι αντιπροσωπείε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μα ενημερώσουν για τα βήματα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί προ την κατεύθυνση αυτή. Και εδώ ε, οι έχοντες την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασχοληθούν με αυτό για να δουν την εφαρμογή, την πρακτική για τις γυναίκες που είναι θύματα βίας και με ερωτήσεις, αναλύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θεωρηθεί απαραίτητο. Και η Ισπανία τώρα που είναι στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσπαθεί πάντα τα θέματα ε, για τις διαφορές μεταξύ των φύλων και τη βία κατά των γυναικών όλα αυτά να συμπεριληφθούν στους συζητήσεις ε, και στι διαπραγματεύσει με τρίτε χώρες από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό και στα πλαίσια του διαλόγου ας πούμε μεταξύ Μολδαβίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης που χθε ε, διεξήχθη στο Τσισινάου στο διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας ε, αύριο την Παρασκευή στην Γενέβη. Και ακόμα επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέχει ώστε εκεί όπου αντιμετωπίζουμε παρόμοια θέματα που έχουν να κάνουν με τη βία κατά των γυναικών όλα αυτά συμπεριληφθούν και να αναφέρονται εκεί μορφές διακρίσης ή βίας. Και επίσης στα πλαίσια ε, συμφωνίας με το Μεξικό, να δούμε το μηχανισμό για να δούμε την, αν πραγματικά ισχύει η νομοθεσία κατά το γυναικών. Και θα πρέπει η πρωτοβουλία αυτή να προωθηθεί και πάλι στην επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ισπανία, έχοντας την Προεδρία, επίση έχει συμπεριλάβει στην μέση διάταξη ένα σημείο που αφορά την βία κατά των γυναικών και συγκεκριμένα κατά το τρομερό αυτό έγκλημα ε, η θανάτωση γυναικών και στο Κοχόμ 12 και 13 Απριλίου που θα λάβει χώρα αυτή η συνάντηση θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη βία κατά των γυναικών και τις διακρίσεις ε, ανάμεσα στα δύο φύλλα και ακόμα κάτι όλα αυτά που κάνει η Ισπανία έχοντας την Προεδρία θα προσπαθήσουμε Τώρα, 10 χρόνια μετά από τις αποφάσεις ε, ε, το 13, 25 18, 20 από την, ε, τα Ηνωμένα Έθνη. Εδώ όλα αυτά είναι μόνο ένας, ε, μια πτυχή από αυτές τις προσπάθειες. Το αποδείξαμε, το είπαμε από τα χειρότερα που έχουν γίνει και πραγματικά η εθνική συμφιλίωση μετά από εχθροπραξίες, από ένοπλη σύραξη απειλείται εάν συνεχίσουν να ισχύουν αυτά και ακόμα το 1325 και 1820 και 1325 ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν στα, στα πλαίσια της ε, πολιτικής, ε, εξωτερικής πολιτικής. Εδώ στα πλαίσια όλα αυτά θα πρέπει να δούμε για την εφαρμογή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτών των ε, ψηφισμάτων και των ψηφισμάτων στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Επίσης ε, μέσα οικονομικά από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και σύμβουλοι εμπειρογνώμονες για παρόμοια θέματα παντού σε όλες τις αντιπροσωπείες πολιτικές στρατιωτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα προγράμματα δράσης εθνικά για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 η Ισπανία είναι από τα 16 κράτη των Ηνωμένων Εθνών και από τα 9 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προώθησαν παρόμοιο πρόγραμμα και σχέδιο. Ε, και άλλοι ε, επίσης ε, άλλοι τρεις προωθούν παρόμοια σχέδια με Γενικό Γραμματέα ασχολούμεθα, εξετάζουμε το θέμα αυτό και υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Γι' αυτό ακριβώς η Ισπανία έχει προτείνει διάφορα συγκεκριμένα μέτρα για ενδετικοποίηση της μάχης αυτής και μια εφαρμογή αυτών των ψηφισμάτων. Εδώ θα αναφέρουμε ορισμένα όπως είναι η συνεργασία με τη Βελική επόμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 χρόνια μετά από την υιοθέτηση του 1325 και επίσης 24 Μαρτίου στη Μαδρίτη ένα σεμινάριο από το Υπουργείο Άμυνας για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 στα πλαίσια της ε, και στα ΚΕΠΑ και στα κράτη-μέλη και με την Εσθονία που θα ασχοληθεί με τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής και την εφαρμογή στα πλαίσια του ΝΑΤΟ μια έκθεση με συστάσεις πρακτικές που θα αφορούν το μέλλον και επίσης θα πρέπει να αναφέρομαι τη συμφωνία για ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η εφαρμογή της ψηφίου 1325 εργασίες στα τελικά πλαίσια του Peace Building Commission της Επιτροπής Οικοδομής Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών. Ολοκληρώνοντα, έχοντα την Προεδρία εμεί η Ισπανία, συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τον αγώνα αυτό κατά τη διάκριση των φύλων και κατά τη βία των γυναικών. Είναι από του κύριου τομεί με προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη στο θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό επειδή αυτό το πρόβλημα όλο και γιγαντώνεται, αλλά για να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθειά μα, όλο και περισσότερε κυβερνήσει καταλαβαίνουν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και ότι η απειλή τη παραδόσεις τους και οικονομικά και κοινωνικά τους απειλεί επίσης. Και κάθε φορά περισσότερες κυβερνήσεις έχουν διάθεση πραγματικά να συνεργαστούν για να ε, μην υπάρχει πια αυτό πρόβλημα και από την κοινωνία των πολιτών και από παντού που δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση αυτή. Η, πρόκλησή μας τώρα είναι να καταλάβουν όλοι την, πόσο δεινό είναι το πρόβλημα μέσω εκστατιών ευαισθητοποίηση και προ τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα και ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να είναι κάτι το θεσμοποιημένο στην κοινωνία η βία αυτή. Και επίση η μάχη κατά τη βία κατά των γυναικών θα πρέπει να παραβάνει όλε τι πτυχέ με πολλαπλέ λύσει πρόληψη, στήριξη στα θύματα όπω επίση και τιμωρία των εγκληματιών. Και αυτό, αυτό θα πρέπει να ισχύσει σε όλες τις κοινωνίες ολόκληρου του κόσμου. Ευχαριστώ. Thank you. And... Uh, Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βερονίκα, Αρνό, Διευθύντρια της ε, Γενικής Διεύθυνσης Δημερών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να πληρώσω όσα είπαν οι προηγούμενοι και μάλιστα ταπεινά ταπεινά. Ε, ε, ευτυχώς είμαστε μακρύ πολύ πιο μακριά από εκεί που σημαίνεται αυτή η βία, τουλάχιστον σε σχέση με την εκπρόσωπο του Κόγκο. Εδώ το Κοινοβούλιο πολύ σωστά επικεντρώνεται στο πρόβλημα αυτό, γιατί έχουμε το ψήφισμα αυτό αυτό 13-25, 10 χρόνια μετά. Είναι κάτι το σημαντικό, την πρώτη φορά ακριβώς που το Συμβούλιο Ασφαλείας έδειχνε καθαρά πως έχει βία στις ένοπλες σειράξεις, η βία κατά των γυναικών, το είπαν και οι συνάδελφοι, και ήταν ένα μέσο με στα πλαίσια ενός πολέμου όπως όλα τα υπόλοιπα. Δέκα χρόνια λοιπόν μετά και από αυτά που προσπάθησε να κάνει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το έκανε και ο Γενικός Γραμματέας των Εθνών, είναι ε, ο κ. Μουν είναι να δοθεί ακριβώ προσοχή σε αυτό και όχι έτσι προχείρα, αλλά χρειάζεται συγκεκριμένη πρόοδο και προ στιγμή να σα πω ότι ανησυχώ για αυτό το γεγονό ότι σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών τα πράγματα δεν είναι κατάλληλα οργανωσμένα όπω πρέπει τουλάχιστον και κάπω καθυστερούμε στι όλε συζητήσει για το θέμα αυτό, έστω και αν εκδηλώνεται ιδιαίτερη πολιτική βούληση. Σημαίνεται μια κάποια πρόοδο, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη χρονιά αυτή και τον Εύρο που μα πέρασε στα Ηνωμένα Έθνη. Για πρώτη φορά τα Ηνωμένα Έθνη ακριβώ μετά από μια συζήτηση για το θέμα του Κονγκό υιοθέτησαν ένα πρόγραμμα κατά τη βία εναντίον των γυναικών στα πλαίσια ενόπλων σειράξεων και με κυρώσει παρακολούθηση, έλεγχο και τώρα γνωρίζουμε ότι ε, από πλώς επιτρόπου Ολστρομπ ε, ε, γίνεται ένα έλεγχο. για και έρευνα και στη Γενέβη επίσης ε, στο Συμβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα συζητήθηκε το Κονγκό αλλά όχι μόνο για περιπτώσεις ακριβώς ε, παραβιάσεων παρομοίων και όπως είπε συνάδελφος από την Ισπανία είχαμε και παρόμοιες αναφόρες ε, για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προληπτικά και προσπαθούμε να πούμε ότι υπάρχουν στη διάθεσή μας διάφορα μέσα και ένα από τα προβλήματα είναι όλα αυτά να μπουν σε κοινή βάση και από στατικής πλευράς και από κοινωνικής πλευράς πέρα από τα παραδοσιακά όπως το είπε η συναδελφός, ε, βέβαια δύσκολο είναι ανάμεσα στα κατεπήγοντα μέτρα και στα μη κατεπήγοντα να κάνουμε μια διάκριση και ανάμεσα στα πολιτικά και στα στρατιωτικά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι κάπως να συντονίσουμε την όλη κατάσταση και πραγματοποιούνται τακτικά συζητήσεις με τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των σχεδίων δράσης. Η Ζανίν είπε ότι το Μπουρούντι και η Ρουάντα διαθέτουν προγράμματα δράσης με εκπλήσει και μάλιστα θετικά αυτό στα 17 κράτη που έχουν παρόμοια, ε, διαθέτουν παρόμοια προγράμματα. Ευτυχώ ή δυστυχώς είναι ευρωπαϊκά και η Λιβερία, η Σιερα πιο άλλο κράτο, άλλο ανακράτο. Α, ναι, και του διαθέτουν πρόγραμμα και χρειάζεται πολλή προσπάθεια. Δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό χρημάτων, είναι και συνήθεια, σας το πούμε έτσι, και διάθεσης βούλησης πολιτικής. Εντάξει, απέναντι στα θύματα δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, αλλά έχει σημασία γιατί θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και οι στρατιωτικοί για το τι μπορούν να κάνουν. Κάτι ακόμα. Ιδιαίτερα βλέπουμε τη, για την ε, ειρήνη και την ασφάλεια τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Έχουμε 12 κράτη πιλωτικά και με την ε, Κονγκό στα πλαίσια της UNIFEM. Κάτι προσπαθούμε να πετύχουμε λοιπόν και προσπαθούμε επίσης να διαθέτουμε ένα μηχανισμό προειδοποίηση και επίσης να διαθέτουμε δείκτε ακριβέστερου για τι πράξει βία κατά των γυναικών. Επίσης προσπαθούμε από πολιτικής πλευράς η Μπεατρίς ε, από την Ισπανική Προεδρία το έθιξε αυτό. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου και συνεργαζόμαστε με την Αφρικανική Ένωση, αλλά από ό,τι φαίνεται καθαρά κάτι τέτοιο δεν επαρκεί. Σχετικά τώρα με τις ενέργειες από πλευράς πολιτών, ε, πολιτών ε, και όχι στρατιωτικών. Ε, εδώ μετά από εκεί που έχουν συμμετέχει οι ευρωπαϊκές έχουμε επιτόπου εμπειρογνώμονε που ασχολούνται με το όργανο σταθερότητα και έχουμε ακριβώ σχετική ενημέρωση και από το 2012 ακόμα περισσότερο θα συμμετάχει ο κόσμος σε παρόμοιες ενέργειες και ακόμη κάτι για τις ΕΚΟ εδώ υπάρχει ειδική ευαισθητοποίηση και για τα παιδιά επίσης. Ε, κύριε Χάουζερ είπε ότι ε, δεν είναι πρόβλημα των γυναικών των ανδρών ο βιασμός, αλλά υπάρχουν ε, και θύματα γυναίκες και θύματα μικρά κορίτσια και δυστυχώς και αγόρια. Όλο και περισσότερο συναντάται το φαινόμενο αυτό και θα πρέπει να συντονιστούμε και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις υπάρχουν και γυναικών και για τα παιδιά που ασχολούνται και θα πρέπει να σημειωθεί ο απαραίτητο συντονισμός και επίσης ε, στην ΚΕΠΑ, στα πλαίσια της ΚΕΠΑ υπάρχουν επιτόπου σύμβουλοι και στη, στο στο Κωσυφοπέδιο υπάρχουν αυτοί οι σύμβουλοι και να σας πω και κάτι για το Κονγκό ολοκληρώνοντας κάτι που δείχνει καθαρά πόσο περίπλοκο είναι το θέμα και το πρόβλημα. Για να δούμε τι γίνεται να στηρίξουμε τα θύματα ψυχολογικά, με φάρμακα κλπ. Και επίσης να, ε, να αποφύγουμε την ατιμορρησία και στηριζόμαστε και στα ψηφίσματα των Εθνών και ακόμα και αυτό αναφέρθηκε από προηγούμενου συναδέλφους ε, το σχετικό σχέδιο για την ε, απόδοση δικαιοσύνη στις ανατολικές περιοχές και επίσης ε, να δούμε ότι ε, ασχολούνται και με τη σεξουαλική βία πέρα από τις άλλες ε, αρμοδιότητες από το Μάρτιο που μας πέρασε και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία χρηματοδοτούν αυτές τις προσπάθειες και προσπαθούμε να πετύχουμε συντονισμό στα κράτη-μέλη. Και ακόμα κάτι προσπαθούμε να κάνουμε την UNIFEM να δράσουμε προληπτικά. Αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω ότι πρόκειται κάτι, επιτρέψτε μου να το πω, ότι να είναι κάτι το πρότυπο και στο Κοινοβούλιο να ασχοληθούμε με την εξωτερική πολιτική και με το ρόλο των ειδικών αποσταλμένων και θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν περισσότερο και καλύτερα υπόψη και επίσης σημειώθηκαν συζητήσεις στις ομάδες Συμβουλίου και αποστολή διερεύνησης ε, από πλευρά Συμβουλίου και ειδικοί εκπρόσωποι για την περιοχή των Μεγαλολιμνών, ο κ. Ντεγκύρ, για να ελέγξουν το πρόβλημα αυτό της σεξουαλικής βίας θα παραταθεί η εντολή του και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να βοηθήσει η κυρία Μικανιέρβα όπως είπε, θα πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα που έχουν σημασία μεγάλη θα πρέπει επιτόπου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τις αγροτικές περιοχές ε, που δεν υπάρχει μια υποδομή ε, ούτε από υγειονομικής πλευράς ούτε από νομικής πλευράς ε, και επίσης να ακουστούν λοιπόν αυτά τα σχόλια. Είπαν όλοι επίσης ότι απαιτείται ιδιαίτερη αντίδραση. Ποιο είναι το θετικό τώρα. Όλοι παραδέχονται ότι είναι απαράδεκτα παρόμοια εγκλήματα και όχι δοθεί δημοσιότητα και μεμονωμένα όσον αφορά τα θύματα, μια κινητοποίηση και τώρα το 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλοι οι φορείς να μπορέσουν να κινητοποιηθούν κατάλληλα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το παίρνουν σοβαρά ακόμα και στρατιωτικοί και στρατιωτικοί εδώ το επίσης από ευρωπαϊκής πλευράς τι αποστολές το έχουν κατανοήσει αλλά σημαίνει ταυτόχρονα ότι και οι πολίτες θα το θα απασχολήσει περισσότερο ακόμα ε, λοιπόν ε, ε, από τη στιγμή που θα το προσέξουν αυτό θα προσέχουν με περισσότερο συστηματικό τρόπο επίσης ε, από πλευρά αστυνομία ε, θα πρέπει να κατανοήσουμε με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε τοπικό επίπεδο επίσης τις μικροοργανώσεις και αυτό που λυσμό να σας πω για το Κόγκο είναι ότι το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουμε ένα πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτόπου που έχουμε αναπτύξει επιτόπου και έτσι οι μη κυβερνητικές τοπικές οργανώσεις μπορούν περισσότερο να έχουν κάποια κονδύλια για να βοηθηθούν και να βοηθήσουν και περισσότερες επαφές όσο γίνεται επιτόπου με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Είναι βέβαια πολύ μεγάλη χώρα το Κονγκό και δύσκολο είναι να ασχοληθούμε όλα όσα είναι και στην Κινσάσα και στα ανατολικά του Κονγκό να σας πω ότι εκεί χρειάζονται να καταβληθούν ακόμη περισσότερες προσπάθειες με ε, άτομα για επαφή ε, σε θέματα δικαιοσύνης, υγειονομικά, παιδιά, γυναίκες, ε, όλους. Σας ευχαριστώ πάντως για τη δυνατότητα που μας προσφέρετε ώστε από πολιτικής πλευράς να μπορέσουμε να το ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το θέμα. Είναι πολύ σημαντική η χρονιά και μέσα του ψηφίσματος 1325 και από την Αιόρκη και από παντού και με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αυτή την προσέγγιση με κατανόηση και ε, Ηνωμένα Έθνη όλοι αυτοί και ότι έχουμε ε, από τον Γενικό Γραμματολόγο Εθνών ειδικό απεσταλμένο για τα θέματα των γυναικών και άκουσα με προσοχή αυτά που είπαν όσοι συναδελφοί εργάζονται επί τόπου και ε, μας βοηθούν εμάς που είμαστε μακριά από τις χώρες αυτές να μπορέσουμε να τα αντιδράσουμε όσο γίνεται ταχύτερα και καλύτερα. Ευχαριστώ κύριε Αρνό. Θα ήθελα να καλωσορίσω και την πρόεδρό μας, την Χάιρι Χάουτελα. Πολύ χαιρόμαστε που γυρίσατε στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια. Άννα Γκόμες, Λόχμπιλερ και Χάουταλα. Η Άννα Γκόμες πρώτα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ που οργανώσατε αυτό, αυτή την ακρόαση για αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να φύγω αμέσως, όχι γιατί δεν με ενδιαφέρει το ζήτημα, αλλά γιατί πρέπει να πάω στην Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας όπου θα έρθει ο Υπουργός Άμυνας ε, ή Υπουργός Άμυνας μάλιστα της ε, Ισπανίας, οπότε πρέπει να πάω εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Αυτά που γίνονται λοιπόν στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και όπως είπε και ε, η κυρία μου Κανίρουα δεν είναι μοναδικό φαινόμενο, το έχουμε δει και στα Βαλκάνια, το έχουμε δει πολλές φορές ε, γιατί ε, το έγκλημα αυτό συμβαίνει πολύ συχνά και είναι συχνά πολεμικό όπλο. είναι γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα έχου, έχει συχνά παραγνωρίσει το πρόβλημα αυτό και δεν ανασκουμπώνεται για το ζήτημα αυτό. Όλη η δουλειά που έκανε η Ισπανική Προεδρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευαισθητοποίηση, όλη αυτή, ε, όλα αυτά τα λόγια για τα οποία μίλησε η κυρία Αρνό, καλά είναι, αλλά χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα από αυτό. Και είναι γεγονός ότι η κατάσταση στο Κονγκό Επιζητεί επιτέλους λύση. Πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα. Έχει πάρα πολύ επενδύσει πόρους η χώρα. Το πρώτο, η πρώτη ε, αποστολή της ΚΕΠΑ ήταν ε, συγκεκριμένα στο Κονγκό. Μετά το 2008 υπήρχε μια αποστολή για την ε, ασφάλεια στο πλαίσιο των εκλογών πάρα πολλέ αποστολές και της ε, μοστία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δεν βελτιώνονται τα πράγματα. Αντιθέτως γίνονται χειρότερα. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Δεν επικεντρωνόμαστε αρκετά στο πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει ορατότητα, να είναι γνωστό το πρόβλημα και βεβαίω και στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση πρέπει να είναι πιο γνωστό το πρόβλημα αυτό. Ε, και η πρώην ε, Επίτροπος μπορεί να μας βοηθήσει αλλά πρέπει και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσουμε μια πιο συνεπή προσέγγιση, πιο αποτελεσματική προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων μέσων που χρησιμοποιούμε και είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά τέτοιου είδους μέσα και είναι δύσκολο να τα συντονίσουμε, να τα ακόμη και εδώ ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ είμαστε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ακούσαμε και μια σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Ανάπτυξης ε, που είναι υπεύθυνη για την ε, συνεργασία μας το Κονγκό σε σε άλλες πτυχές της, δεν είμαστε πάρα πολύ συντονισμένοι. Πρέπει να συνδεθεί η Επιτροπή Εξωτερικών, η Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας, ε, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Επιτροπή Γυναικών. Μιλάμε για μεγάλο συντονισμό. Εμείς προτείνουμε μια αποστολή προτεραιότητας όχι μόνο στην Κινσάσα, Έχουμε πάει από το 2006 πολλές φορές. Πρέπει να υπάρχει μια αποστολή προτεραιότητα όπου θα μπορούσαμε να πάμε σε αυτές τις ε, περιοχές της υπαίθρου, ε, τις πιο ε, περιφερειακές. Να υπάρχει λοιπόν μια κοινή αποστολή όλων των επιτροπών που είναι αρμόδιες για αυτό το θέμα και βεβαίως να εμπλέξουμε και το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα θέματα της υποστήριξης των θυμάτων, της ατιμορρησίας. Ε, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε την τοπική κοινότητα. Οι γυναίκες δεν είναι μόνο θύματα. Μπορεί να είναι παράγοντες της ειρήνης και της εσφέλειας. Και εφόσον ε, τόσο άσχημα τα έχουν ε, καταφέρει οι άντρες στην περιοχή, νομίζω ότι επιτέλους έχει φτάσει η στιγμή να δώσουμε δυνατότητα και στις γυναίκες να συμμετέχουν. Πάρα πολλές γυναίκες υποψήφιες υπήρχαν στο Κονγκό, δεν εξελέγησαν αν δεν τις υποστηρίξαμε σωστά και γι' αυτό εν μέρη δεν εξελέγησαν, πρέπει ακριβώς να μπορέσουμε να θέσουμε τα πράγματα όλα αυτά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να ζητήσουμε από όλα τα μέσα που αφορούν την αναπτυξιακή ανεργασία, ε, ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα και στις εταιρείε ανάπτυξης που υπάρχουν στο Κονγκό και τις οποίες εμείς προσπαθούμε να υποστηρίξουμε, να λάβουν υπόψη αυτό το θέμα, να τους γνωστοποιήσουμε ότι έχουν και εκείνες οι εταιρείε ε, ευθύνη για την ε, βία τη συνεχιζόμενη κατά των γυναικών. Αν επικεντρωθούμε σε αυτό, μπορούμε να ε, αλλάξουμε την κατάσταση ε, της ασφάλειας στο Κονγκό και μιλάμε για μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου και η ευθύνη για την προστασία και η ασφάλεια και η σταθερότητα μπορούν να συνδεθούν για να υπάρξει κάτι το συγκεκριμένο. Δεν είναι μόνο δηλαδή θεωρία. Μπορούμε να περάσουμε στην πράξη. Επί που μπορούμε να βοηθήσουμε, να κάνουμε τη διαφορά και ελπίζω πραγματικά ε, να είναι μια τέτοια πρωτοβουλία της ε, Επιτροπής μας ε, και να υπάρξει αυτή η αποστολή προτεραιότητας που ανέφερα για να έχουμε συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λόχπιλερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η πρόταση της κυρίας Γκόμες να πάει στο Κονγκό μια μεικτή αντιπροσωπεία πολλών επιτροπών είναι εξαιρετική. Θέλω να ευχαριστήσω όμως και την Ισπανική Προεδρία, διότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα και κάνει διαφοροποιημένες προτάσεις για η δουλειά πρέπει να γίνει κατά της βίας κατά των γυναικών. Και οι προεδρείς που θα ακολουθήσουν, Βουλγαρία και Ουγγαρία, θα πρέπει να αναλάβουν το θέμα, να παραλάβουν τη σκητάλη δηλαδή και να συνεχίσουν, διότι ε, υπάρχουν και συνέπειες στην εφαρμογή. Σεις κύριε Χάουζερ είπατε πόσο σημαντικό είναι να υποστηριχθούν μικρές μη κρατικέ οργανώσεις που δρούν επιτόπου. Η κυρία Αρνό είπε ότι μειώνει για παράδειγμα τα κατόφλια ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν υποστήριξη και οι μικρές μη κρατικές οργανώσεις. Μπορείτε να πείτε με κάπως ακριβέστερο τρόπο με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει πιο εφικτή η ε, χρήση του χρηματοδοτικού αυτού μέσου. Είπατε επίση πόσο σημαντικό είναι να υποστηριχθούν οι υπερασπιστέ των ανθρώπινων δικαιωμάτων που αντιτάσσονται γυναίκες είτε άνδρε κατά της ε, γενετήσια βία, αλλά εκείνοι επίση οι οποίοι τάσσονται και μάχονται υπέρ των δικαιωμάτων γενετησίων και άλλων των ε, ε, προσώπων. Και θα υπάρξει και ιδιαίτερη έκθεση για την προστασία των ε, υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Είμαι βέβαια ότι θα περιληφθεί εδώ στις εργασίες μας. Εμείς εδώ στην υποεπιτροπή μας προκερού, δεν είμαι βέβαια, είχαμε αναθέσει μια μελέτη η οποία επρόκειτο να εξετάσει τι κάνουν οι διάφορες μη κρατικές οργανώσεις, κατά πόσον το ψήφισμα 1325 πραγματικά εφαρμόζεται και στις χώρες μέλη αλλά και εκτός αυτών. Ακούω τώρα πολλούς να επενούν το ψήφισμα αυτό. Βέβαια είναι δύσκολο στην εφαρμογή του. Ίσως πρέπει να σκεφτούμε αν ίσως πρέπει και εμείς να εργαστούμε προς την κατεύθυνση εγκρίσεως ενός ψηφίσματος που θα αναφέρεται σε ελάχιστες προδιαγραφές για την εφαρμογή του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών. <coughs> Ίσως είναι καλό γιατί κλείνει μια δεκαετία από τότε που ψηφίστηκε, τον Οκτώβριο. Να μην είμαστε απλώς ικανοποιημένοι μόνο από το ότι το κράτος κύρωσε το ψήφισμα του ΟΗΕ, το βελγικό υποθέτω ότι εννοεί, μέχρι τώρα 11 χώρες έχουν κυρώσει το ψήφισμα αυτό η δική μου χώρα, η Ομοσπονδιακή Γερμανία, δυστυχώς δεν έχει θεωρήσει ότι πρέπει να ε, εγκρίνει ένα σχέδιο δράσεως το οποίο να συνδεθεί με το ψήφισμα αυτό των Ηνωμένων Εθνών. Ίσως λοιπόν πρέπει, όπως είπα, να συντάξουμε ένα ψήφισμα το οποίο να ε, αναφέρεται στην εφαρμογή του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών. Η κυρία Χάιντι Χαουτάλα. Ευχαριστώ πολύ που με βοηθήσατε στην Προεδρία. Τρεις ώρες καθυστέρηση είχε πτήσει από τη Νέα Υόρκη. Γι' αυτό άργησα. Το ζήτημα αυτό της βίας κατά των γυναικών σε ένοπλες συγκρούσεις με ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι κάτι το οποίο έχει πολλές φορές εξετάσει η Επιτροπή στην οποία συμμετείχα και πρέπει να πω ότι ο Μπάνκι Μουν, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, με πολύ έντονους όρους ε, μίλησε για το θέμα αυτό. Σε πολύ ψηλό επίπεδο λοιπόν ε, εξετάσαμε το ζήτημα αυτό γιατί πρόκειται για πολύ σοβαρό πρόβλημα. Επίσης ε, συνάντησα την Τζέσικα Νάιτον στο γραφείο της στη Νέα Υόρκη και μιλήσαμε για αυτό το θέμα και Είπαμε επίσης ότι το ζήτημα των φίλων θα έπρεπε να αποτελεί τμήμα όλων των συζητήσεων και όλων των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν κάποιες απτές πρόοδοι για τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσπαθήσαμε να δείξουμε πού ακριβώς υπήρξε πρόοδος. Και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν στο επίκεντρο της προσοχής, γιατί Βρισκόμαστε στη δέκατη επέτειο του ψηφίσματος 1325 και αυτό μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να επισπεύσουμε τη διαδικασία. Όμως, δυστυχώς, Μόνο 17 χώρες συμμετείχαν ε, στο πρόγραμμα δράσης. Η Επίτροπος ε, Βάλστρομ είχε περιορισμένη εντολή ως προς το ζήτημα αυτό της ε, βίας κατά των γυναικών σε ένοπλες συγκρούσεις. Ίσως θα έπρεπε όχι μόνο να ασχολούμαστε με το θέμα της βίας κατά των γυναικών σε ένοπλες συγκρούσεις, αλλά και στη συμμετοχή των γυναικών στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να σταματήσουν οι ένοπλες αυτές συγκρούσεις. Να διευρύνουμε δηλαδή ακόμη περισσότερο τη συζήτησή μας. Δεν πρέπει να συνεχιστεί η ατιμορρησία, δεν πρέπει καθόλου να απομακρύνουμε την προσοχή από το θέμα αυτό. Ως προς το ψήφιμα 1325 πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο και ενδεχομένως να χρειαστεί και ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να θέλει να πάρει το λόγο. Οπότε, στρέφομαι προς τους ομιλητές μας τους προσκεκλημένους μας ε, αν θέλουν να πάρουν το λόγο και να σχολιάσουν αυτά που άκουσαν από τους συναδέλφους και θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε όσο το δυνατόν συντομότεροι γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα στην ημερήσια διάταξη. Η Δόκτωρ Χάουζερ. Θα απαντήσω στα γερμανικά και, και θα προσπαθήσω να είμαι και σύντομη βέβαια. Ε, είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξω ξανά τα όσα είπε η Ζανίν εδώ αριστερά μου, ε, ότι δηλαδή γυναίκες υποψήφιες πρέπει να υποστηρίζονται. Υπάρχουν πολλοί ικανές γυναίκες πολιτικής στο Κονγκό και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προσκαλέσει τις γυναίκες αυτές εδώ στις Βρυξέλλες να καταστήσει τις αφές ότι τις θεωρεί ικανές και να δώσει και ένα μήνυμα με τον τρόπο αυτό. Ότι δηλαδή τους προσφέρει ε, αναφανθόν υποστήριξη. Συνεργασία με τις μικρές, ε, μικρές ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Εγώ το λέω και το ξαναλέω αυτό. Ακούω και από την κυρία Αρνό αλλά και από την κυρία της Ισπανικής Προεδρίας διάφορες προτάσεις. Εγώ θα χαρώ πάντως ιδιαίτερα εάν εν ευθέτω χρόνο μπορέσουμε να ξαναειδωθούμε, να συζητήσουμε συγκεκριμένα δηλαδή για τα ποια πράγματα μπόρεσαν να εφαρμοστούν, ποια όχι και γιατί. Και σας παρακαλώ πραγματικά έντονα πράγματα τα οποία γράφονται στα χαρτιά δεν συμβαίνουν επί τόπου όμως. Οι ντόπιε γυναικείς οργανώσεις ας προσκληθούν εδώ ως εμπειρογνώμονες για όλα τα πράγματα που αναλαμβάνετε εσείς εδώ. Σημαντικό είναι επίσης να πω ότι είναι σωστό να ε, θεσπιστούν μίνιμουμ προδιαγραφές για την εφαρμογή. Νομίζω ότι αυτό άλλωστε είναι και το βασικό πρόβλημα. Στα χαρτιά τα έχουμε γράψει όλα όσα χρειάζονται, ήδη από το Πεκίνο, με ψηφίσματα. Αλλά τι ωφελεί, τι ωφελούν τα λόγια της γυναίκης επιτόπου εάν δεν, δεν ελέγχουμε την εφαρμογή. Το πώς ασκείται η δικαιοσύνη σε καθημερινή βάση, πώς ε, λειτουργεί η αστυνομία σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό λοιπόν ο έλεγχος και η παρακολούθηση, το monitoring είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Θα τονίσω και πάλι την αξίωση που προέβαλα πριν την ε, θέσπιση της θέσης μιας ειδική εκπροσώπου για το πρόβλημα αυτό, η οποία να μπορεί να αναλάβει στα χέρια της τα ενία πολλών δραστηριοτήτων, γιατί είναι σημαντική η διαδικασία αυτή, πολύ σημαντική ώστε να αφαιθεί μοναχά στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι έχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα να χειριστούν όπως το διαπίστωσα πάλι εδώ σήμερα. Χρειάζεται λοιπόν να μπορεί το πρόσωπο αυτό να αναλάβει δράση συγκεκριμένα. Βλέπω ότι είναι εξαιρετικές οι προθέσεις σας, αλλά χρειάζεται όπως είπα ανάληψη δράσης συγκεκριμένης. Εν τέλει εκφράζω τη λύπη μου, διότι έχουμε μόνο 11 ε, σχέδιο δράσης εδώ. Μα δεν έχουμε 11 σχέδια δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λυπηρό από πλευρά ε, Ομοσπονδιακή Γερμανία ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί απαραίτητο να θεσπιστεί ένα γερμανικό εθνικό σχέδιο δράσης και ιδίω εν του γεγονότος ότι και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφεύγουν ατιμωρητοί. Ο πρόεδρος του FTLR του FDLA στην Γερμανία που δρούσε επί χρόνια ως ε, πρόσωπο που, ε, που έχερε ασύλου στη Γερμανία και όμως μπόρεσε και με τον τρόπο αυτό και κινούμενος ελεύθερος στη Γερμανία, ε, ελεύθερος στη Γερμανία να οργανώσει διάφορες φαγές στο Κονγκό. Το ίδιο και αλλού και στη Γαλλία έχουν, υπάρχουν τέτοια πρόσωπα και στο Βέλγιο και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν πολλές και περίπλοκες ε, αρμοδιότητες και ε, διασυνδέσεις όπου πρέπει κάποιος να καθίσει να τα πάρει αυτά τα πράγματα, να τα εξετάσει αυτά τα πράγματα όλα μαζί. Μιλήσατε επίσης και για την U4 όπου υπήρχαν gender advisors, δηλαδή σύμβουλοι ειδικά για τα θέματα ισοτιμίας των φύλων. Εμείς ε, είμαστε σε στενή επαφή με την Charlotte Isaacson ε, Σουηδή σύμβουλο για θέματα ε, ισότητας των φύλων καθημερινά άκουγε παράπονα και καταγγελίες, καταγγελίες από ε, γυναίκες στρατιωτικούς διεθνών στρατιωτικών σωμάτων που πήγαιναν εκεί και παραπονούνταν και για σεξουαλική παρενόχληση από τους ανωτέρους τους ή από άλλους συναδέλφους τους και δεν είχαν συνομιλητή για να απευθυνθούν. Χρειαζόμαστε λοιπόν εδώ και αυτό. Φανταστείτε δε πόσο περισσότερο τις ε, γυναίκες και τα κορίτσια του Κονγκό που δεν έχουν απολύτως κανέναν για να απευθυνθούν και να καταγγείλουν. Όταν για παράδειγμα υφίστανται βιασμούς από ε, προσωπικό των διεθνών στρατιωτικών δυνάμεων που εδρεύουν επί τόπου ή και από πολιτικό προσωπικό των δυνάμεων αυτών. Η κυρία Ισαξον ήταν η μοναδική αξιωματούχος εκεί επιτόπου η οποία δεν είχε κάποιον συνομιλητή αντίστοιχα εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ κυρία Χάουζερ. Εσείς κυρία μου. Πολλά πολλά ευχαριστώ και ευχαριστώ για όλα τα σχόλια, τα θετικά σχετικά με την εργασία της ε, Ισπανικής Προεδρίας. για τα σχόλια της κυρίας Γκόμες για μια συνοχή σε όλες τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μάχη κατά του προβλήματος αυτού και την επιτόπου παρουσία και την πρόταση μιας κοινή αποστολής στο Κονγκό που θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε είδαμε ότι απαιτείται κάτι τέτοιο σαν Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να προωθήσουμε και τη σύνταξη τοπικών, την ε, τοπικών στρατηγικών από τις πρεσβείες των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επιτόπου φορείς και είναι σε στενή επαφή με την κοινωνία των πολιτών και είναι στην καλύτερη δυνατή θέση για να έχουν μια συνολική εικόνα όλων αυτών που υπάρχουν, ποια λειτουργούν, ποια όχι, πώς θα ολοκληρωθούν αυτά, πώς θα προωθηθούν και πώς θα έχουμε συγκεκριμένε ενέργειες πάνω σε αυτή τη βάση οι τοπικές στρατηγικές και ελπίζω, ελπίζω ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν για καλύτερη συνοχή επιτόπου για τα σχόλια της κυρίας Λοχπύρα και το ότι οι ενέργειες μας και οι προτεραιότητες μας θα διαρκέσουν και από το Βέλγιο και την Ουγγαρία τις επόμενες προεδρίες ελπίζουμε είμαστε στη στενή επαφή και με τους Ούγγρους και με τους Βέλγους για τη συνέχιση των ενεργειών για τις προτεραιότητες αυτές τοπικές στρατηγικές που έχουν ε, μια θέση μέχρι το 2012 τουλάχιστον. Άρα λοιπόν ε, και τόπου αλλά και το προσωπικό στις πρεσβείες ε, που αλλάζει όλα αυτά τα χρόνια θα χαρακτηρίσουν μια συνέχιση των ενεργειών τους και να προωθήσουν την ισότητα των φύλων και τη μάχη εναντίον στη βία κατά των γυναικών και σε να δεν θα είναι μόνο δική μας προτεραιότητα της Ισπανίας αλλά και όλης τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι ένας άξονας που θα ε, διαπερνά χρονικά και επίσης ε, από πλευράς του υπατορμοστή και ακόμα για την, ε, το ψήφισμα για τα ελάχιστα που θα πρέπει να ισχύουν ε, για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 θα είναι μια σημαντική ίσως ιδέα αλλά ταυτόχρονα πολλά έχουμε ξεκινήσει για τη σύνταξη των ελάχιστων προτύπων και κύριε, το είπε, η UNIFEM προωθεί επίσης που κάνει αυτή την ανάλυση συντάσσει δείκτες γενικούς που δείχνουν που μπορούν να είναι χαρακτηριστικοί της όλης προσπάθειας για το πώς μπορεί να εξεταστεί η εφαρμογή του 1325 ψηφίσματος των ΗΕ. ΕΕ. Τα αποτελέσματα και οι δείκτες αυτοί θα ε, έχουμε τον Απρίλιο στις Ηνωμένα Έθνη φέτος και πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον θα ήταν να τα δούμε τα αποτελέσματα όλα αυτά. Εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχουμε ένεργα επίσης και να δούμε τι άλλα μέσα εργαλεία θα απαιτηθούν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αρνό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε η εκπρόσωπος της Ισπανικής Προεδρίας για την UNIFEM. Συνεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα αποστελεί ένα ερωτηματολόγιο στις 18 αποστολές ε, και πά της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα ενόπλων συγκρούσεων και της κατάστασης μετά τις ε, ενόπλες συγκρούσεις, όπως είπε η Μπεαντρίς, για να καταρτήσουμε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το θέμα αυτό όσον αφορά την πολύ περιορισμένη εντολή της ε, ειδική εκπροσώπου των, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αυτή ήταν πάντοτε η θέση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάντοτε θέλαμε να διευρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εντολή πρέπει όμως καταρχάς να συνεργαστούμε, με τα, να συνεργαστούμε βάσει των μέσων που έχουμε και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να τα διευρύνουμε. Αυτή είναι η άποψή μας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Τσιπάμπου. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα σε σχέση με την εφαρμογή των ε, προγραμμάτων ε, δράσης ε, του ψηφίσματος 1325. Υπάρχουν πολλά τέτοιου είδους προγράμματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στη Ρουάντα και στο Μπουρούντι με σκοπό ακριβώς να υπάρχει ένα περιφερειακό πρόγραμμα εφαρμογής. Επειδή η περιοχή των μεγάλων ε, λιμνών δεν περιορίζεται πια σε αυτές ε, τις τρεις ε, χώρες μόνο, δηλαδή είπαμε ότι δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε ένα ενδοπεριφερειακό, να έχουμε ένα ενδοπεριφερειακό πρόγραμμα, δηλαδή μεταξύ της περιοχής των ε, ε, μεγάλων ε, λιμνών και 11 χωρών. όμως όλες οι χώρες που είναι μέλη του προγράμματος αυτού θα έπρεπε να συνεργαστούν πριν να υπάρξει ένα πρόγραμμα εφαρμογής ε, Ρουάντα, Ουγκάντα, Μπουρούντι, ε, Τανζανία, ε, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αγγόλα, η Κεντρική Αφρική, το Σουδάν. Και υπάρχει και μια χώρα που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία ήδη επεξεργασίας ε, του περιφερειακού προγράμματος εφαρμογής, γιατί ακριβώς οι μελέτες έδειξαν ότι το ψήφισμα αυτό δεν εφαρμόζεται στην περιοχή των μεγάλων λιμνών. Αυτά τα προγράμματα υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται επαρκώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, ομιλητές μας και τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση. Τώρα, κάποια σχόλια σε σχέση με την ε, συνέχιση ε, της διαδικασίας. Είπαμε ότι είναι η δέκατη επέτειος ε, του ψηφίσματος 1325 από την έγκριση της. Υπάρχει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν του ψηφίσματος 1325 και κατευθυντήριες γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συγκεκριμένα για τις γυναίκες ένοπλες συγκρούσεις και επομένω θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα όταν θα παρουσιαστεί πριν από το Σεπτέμβρη. Όσον αφορά τώρα τους οικονομικούς πόρους και τα μέσα σταθερότητας, ε, συμμετείχαμε στην, ε, στις εργασίες ε, της συνεκτικής προσέγγισης που ανέφεραν πολλοί ομιλητές. Σε κάποια από τα έγγραφα, μία έκθεση για τις αποστολές και πάω στο Κονγκό αναφέρεται ότι δεν υπάρχει γραμμή προϋπολογισμού για την βελτίωση της ενσωμάτωσης της διάστασης ισότητας των φύλων Λοιπόν, ε, Στι ε, δραστηριότητες για το θέμα αυτό που λαμβάνουν χώρα σε τοπικό επίπεδο και οι δράσεις αυτές ε, χρίζουν επιπλέον, επιπλέον απόδοσης πόρων από τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα του μέσου σταθερότητα, μέσων σταθερότητας, υπάρχει ομάδα εργασίας με σκοπό την επεξεργασία του ζητήματος αυτού. Τρίτον, Όσον αφορά την ε, ειδικότερη κατάσταση της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό, πρέπει να είναι σαφής προτεραιότητα στο πλαίσιο των ε, εγγράφων στρατηγικής ε, των χωρών και επίσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι θα γίνουν εκλογές φέτος στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και ε, θα επανέλθουμε για την παρακολούθηση της ε, κατάστασης ε, στη χώρα σε μεταγενέστερο στάδιο φέτος. Αυτά για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξής μας. Να περάσουμε... Στο επόμενο σημείο, που είναι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συγγήτριά μα είναι η πρόεδρος της επιτροπής. η Χάιντι Χάουταλα. Αρμόδια καθήλυνα επιτροπή, επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεση. Κύριε Χάουταλα, έχετε το λόγο. Thank you very much, uh, Chair. Ευχαριστώ πολύ. Το έγγραφο ε, ελπίζω να το έχετε μπροστά σας και στην γλώσσα σας. Είναι περίπου το έγγραφο που είχαμε παρουσιάσει ως έγγραφο εργασίας ε, την συνεδρίαση, συνεδρίασή μας στον Ιανουάριο, αν θυμάμαι καλά. Τώρα έχετε μπροστά σας τις συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες έχω ενσωματώσει στην έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συμβολή πολλών παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών. Ε, χαίρομαι επίσης όλος ιδιαίτερος που η Ισπανική Προεδρία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ε, προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βλέπω επίσης ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται να ε, συνεργαστεί πιο συντονισμένα με το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Ελπίζω λοιπόν ότι οι προτάσεις που έχουμε συμπεριλάβει στην έκθεση να ε, τύχουν ιδιαίτερη αποδοχή ε, ώστε να μπορέσουν ε, να εγκριθούν και να εφαρμοστούν. Βέβαια, αυτό είναι ένα σχέδιο έκθεση. Υπάρχει ακόμη χρόνο για την επεξεργασία του και για την ενσωμάτωση νέων ιδεών. Το πρώτο τμήμα, λοιπόν, αφορά τις, ικανό, τις δυνατότητες στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας και ήδη βλέπετε ότι Ορισμένες από τις προτάσεις ε, απευθύνονται προς την ε, ε, υπατή εκπρόσωπο. Γνωρίζετε ήδη ότι προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλούς τομείς. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστεί ότι θα ενσωματωθούν σε όλες τις πολιτικές και επίσης πρέπει να γίνεται παρακολούθηση ε, βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών ε, που ενέκρινε ε, και αναθεώρησε προσφάτως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα εφαρμογής. Έχουμε πολύ σημαντικές δεσμεύσεις αλλά δεν εφαρμόζονται πάντοτε σωστά και αυτό είναι το πρόβλημα. Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, πρέπει να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους ε, στους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο σημείο 7... Υπάρχει έκκληση της Ισπανικής Προεδρίας για την ύπαρξη ενός ε, τοπικού σημείου επαφής ε, των ε, υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί ως τώρα. Οι προτάσεις δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη συνεπούς και συνεκτικής προσέγγισης στο πλαίσιο της, των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, υπάρχουν προτάσεις για τακτικές ετήσιες συνεδριάσεις μεταξύ περασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διπλωματών που θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλός τρόπος όχι μόνο να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τους διπλωμάτες ε, επιτόπου για τις υποχρεώσεις τους και την ανάγκη συνεργασίας με τους ε, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά θα δημιουργήσει και μια δίωδο στους υπερασπιστές να ε, συνομιλήσουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε της ε, σημασία των γυναικών υπερασπιστών των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πολλές φορές ε, κινδυνεύουν στο πλαίσιο της πολύ σημαντικής δουλειάς τους. Επίσης αναφορά στον, στη βελτίωση του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλά μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο αυτό και πολλά μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα πράγματι συμβαίνει και πράγματι λαμβάνεται υπόψη ε, σε διάφορες ε, συζητήσεις ε, και σε συνόδους κορυφής αλλά και σε διαπραγματεύσεις συμφωνιών Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Επίσης, τονίζουμε την ανάγκη ανεξάρτητων οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών που πρέπει να συμμετέχουν στα ζητήματα, στο διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικαιωμάτων και επίσης ε, εξακολουθούμε να διαφωτίζουμε συγκεκριμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και παρενόχληση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη δουλειά τους. Στη παράγραφο 17, για παράδειγμα, λέμε ότι η δημοσιοποίηση των ονομάτων θα βελτιώσει τον αντίκτυπο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αυξήσει την προσοχή του κοινού συγκεκριμένες περιπτώσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και έχω πλήρη γνώση του γεγονότος ότι ενδεχομένως να είναι προβληματικό σε μερικές περιπτώσεις. Υπάρχει, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η δημοσιότητα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Μερικές φορές κάποιος πρέπει να είναι πιο διακριτικός και να σκεφτεί τους κινδύνους που μπορεί να επιφέρει η δημοσιοποίηση των ονομάτων στους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. εμείς εξακολουθούμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να προσπαθούμε να διευκολύνουμε με άμεση υποστήριξη τη δουλειά των υπερασπαστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η τρίτη κατηγορία προτάσεων έχει να κάνει με τη διαφάνεια και την ορατότητα ως μέτρο προστασίας. Ε, ήδη μίλησα για το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που μπορεί μερικές φορές να είναι χρήσιμο για την ε, δημοσιοποίηση των ονομάτων των ανθρώπων αυτών. Πολλές φορές μια τέτοιου είδους ορατότητα, ε, δημοσιότητα της δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ε, υπερασπιστών αυτών μπορεί να είναι ένα πολύ καλό μέτρο προστασίας. Μία ακόμη έκκληση προς την ύπατη εκπρόσωπο για συστηματικές ε, συναντήσεις με υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ταξιδεύει επίσημα σε τρίτες χώρες. Ε, υποθέτω ότι συμφωνούμε όλοι στην έκκληση αυτή, γιατί Καταλαβαίνω ότι ακόμη διαμορφώνεται η υπηρεσία της ΥΠΑ εκπροσώπου και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ευθύς εξ αρχής ε, να ε, αναμένουμε πραγματική παρακολούθηση της κατάστασης των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τα επίσημα ταξίδια. Επίσης, μιλούμε για το βραβείο Ζαχάροφ, ε, το δίκτυο του βραβείου Ζαχάροφ που δρομολογήθηκε το Δεκέμβριο του 2008, κάτι το οποίο επίσης μπορεί να βοηθήσει το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η τελευταία κατηγορία προτάσεων από την παράγραφο 13 και εξή αφορά την ανάγκη συντονισμένης ε, δράσης, ε, προσανατολισμένης προς τα αποτελέσματα. Και επίσης, μία στο εγχειρίδιο για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση χορηγηθισών θεωρήσεων, που θα μπορούσε να βοηθά τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν πρέπει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να φύγουν από τη χώρα τους. Ε, θα ήθελα να ζητήσω μια συνεδρίαση με, τα, με τους εκπροσώπους των κρατών μελών για τα θέματα αυτά. Αυτό δεν το έχω συμπεριλάβει στο κείμενο. Για να συζητήσουμε τις ε, δυνατότητες βελτίωσης ε, των διαδικασιών χορήγησης θεωρήσεων για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην παράγραφο 26... Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Τσεχικής Προεδρίας για τις πόλεις καταφύγια που υποδέχονται τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους δίνουν προστασία προσωρινή και τους δίνουν τη δυνατότητα να μιλήσουν ε, ε, στους πολίτες. Μπορούμε λοιπόν, ε, διατυπώνοντας την έκθεση αυτή, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε περισσότερο τις προτάσεις της Τσεχικής Προεδρίας. Είχαμε μια ακρόαση τον Ιανουάριο, στην οποία προέκυψε ότι ένα, μία από τις βασικές πρωτοβουλιε δεν γνώριζε αυτή την πρωτοβουλία της Τσεχικής Νοεμβρίας, ε, Προεδρίας. Νομίζω ότι είναι μία πρωτοβουλία που βοηθά καλύτερα στο συντονισμό. Και θα ήθελα να τονίσω επίσης την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ευρωπαϊκών ε, οργανισμών ε, και διεθνών οργανισμών, γιατί δεν ε, ασχολείται μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση με την προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και το Συμβούλιο της Ευρώπης και πληθώρα ε, πρωτοβουλειών ε, της κοινωνίας των πολιτών υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω αυτά είχα να πω σε γενικές γραμμές. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για την κάθε πρόταση, αλλά... Περιμένω εναγωνίως να ακούσω τα σχόλια και των ε, σκιωδών εισηγητών και των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ και εγώ, αγαπητή κυρία Πρόεδρε. οι σκιώδεις ηγητέ των πολιτικών ομάδων. Λάσλο, Βιτόριο Πρόντι, που είναι απόντες. Ο Πρόντι ήταν παρόν στην αρχή. Όμως, έχει αφήσει εδώ κάποιες σημειώσει γραπτός Μαρία Σάλκετ, της φιλελεύθερης, της ομάδας των φιλελευθέρων δηλαδή. Θέλετε να μιλήσετε. Σε αυτό το μεταξύ εγώ θα απευθύνω το καλό ορίσατε στην αντιπροσωπεία των ε, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Euromed, του δικτύου ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Euromed. Δύο εκπρόσωποι είναι παρόντες. Ο κύριος Τρίσελ Ελγιασαμή, πρόεδρος του Ιδρύματος Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Ευρωμέντ και ο κύριος Καμάρης που εκπροσωπεί επίσης το δίκτυο Ευρωμέντ. Αν θα θέλατε να λάβετε τον λόγο, πολύ ευχαρίστως. Ορίστε. Εσείς κύριε Καμάρη. Α, όχι, ο κύριος Ντρίς Ελγιασεμή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Κύριε Συγγήτρια, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα σε ευχαριστήσω γιατί έτσι σήμερα μπορούμε να χάσουμε την απόψή μα για την παρουσίαση αυτή τη έκθεση. Τη θεωρούμε σαν στρατηγική σημασία. Ε, μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνα ακριβώς ε, και να σας πω ότι τα συγχαρητήριά μου για την ποιότητα αυτής της έκθεσης πρόεδρος του Ιδρύματος του Μεσογειακού προσπίζοντας ανθρώπινα δικαιώματα με που σήμερα είναι ανεξάρτητος φορέας και ουσιαστικά ένα ίδρυμα οικονομικής στήριξης ε, και μόνο για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κατεπίγωση καταστάσεις, περιπτώσεις που δεν έχουν δυνατότητα να έχουν χρηματοδότηση για διάφορους λόγους που αναλύονται στην έκθεση και που εργάζονται σε θέματα επίσης λεπτά, ε, το προσωπικό δικαιώματα μεμονωμένα ατομικά. Λοιπόν, συμπληρωματική η δράση μας ε, σε σχέση με τις διεθνείς ενέργειες ε, εμείς ε, απλά και μόνο δεν υπερασπίζουμε αλλά απλά και μόνο υποστηρίζουμε οικονομικά. Πρώτα απ' όλα, οικονομικά λοιπόν ενεργούμε και επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με τους συναδέλφους εδώ υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με πείρα που είναι πάνω από 25 χρόνια και υπερασπίζονται στην περιοχή αυτή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Ανρή Μαγκαλή στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική ήταν στην Amnesty International, στο Human Rights Watch και σήμερα είναι υπεύθυνο στον ίδιο γεωγραφικό τομέα και μάλιστα ε, στον αρμόδιο τομέα. Εδώ λοιπόν θα σας πω για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα επίσης ε, των παρεμβάσεων μας των οικονομικών και επίσης ε, για την οικονομική βοήθεια στα πλαίσια μιας ενίσχυσης των ε, δυνατοτήτων ακριβώς των συνεργατών μας με τέσσερις κύριες με προτεραιότητα χώρες Αλγερία, Τινησία, Αίγυπτο, Συρία, τέσσερις χώρες και η κυρία Ατάλα θα επισκεφτεί προσεχώς. Επίσης, εμείς έχουμε δράσει υπέρ υπερασπιστών ε, για 2,5 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότησή μας είναι μέρη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα σε πολλές ε, συναντήσεις, ε, πολλές συναντήσεις έγιναν χάρη στη δική μας στήριξη και με τη δημοσιεύθηκαν ε, όλα αυτά χάρη επίσης στις μας, τη δική μας οικονομική στήριξη και για αρκετές περιπτώσεις είχαμε βοήθεια ιατρική και σε οικογένειες βοήθεια που προσφέραμε ο Μέσορ Μαλέκ θα κάνει ακριβώς διάφορα σχόλια εκ όλων αυτών και να σας πω ότι είναι στην κατάλληλη θέση για να τα πει όλα αυτά γιατί πριν από δέκα μέρες στην την η αστυνομία περικύκλωσε την οικία του και κανείς δεν μπορούσε να πάει στο σπίτι αυτό και μόνο μετά από μια απεργία πείνας και διεθνή κινητοποίηση τότε μόνο μπόρεσε να κυκλοφορήσει ελεύθερα και να έχει ελεύθερη πρόσβαση. Να έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον προηγούμενο μιλητή και φίλο, πρόεδρο, και να σας πω ότι ε, σας δίνουμε συγχαρτήρια για την έκθεση αυτή, την οποία έχουμε μελετήσει είναι πολύ σημαντικό για μας γιατί δεν ε, αγνοούμε διάφορες υποχρεώσεις της πολιτικής των κρατών μελών που δεν είναι κάτι το εύκολο και στην Τινησία είχαμε την Υποεπιτροπή των Δικαιωμάτων Ευρωπαϊκή Ένωση Τινησία. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν για τις προθέσεις του αλλά είναι μια πικρή αλήθεια πραγματικότητα γιατί για την κοινωνία πολιτών και οι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορούν επιδενή να επικοινωνήσουν ε, η Ισπανική Προεδρία τους αγνόησε. Δυστυχώ, λυπάμαι γιατί στη Μαδρίτη μας είχαν υποδεχθεί πολύ ζεστά. Λοιπόν, ε, αυτό είναι αρνητικό. Εδώ θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω, επικεντρώσω την προσοχή μου σε λίγα σημεία. Πρώτα απ' όλα τη σημασία πέρα από την έκθεση, αλλά θα πρέπει να το δείξουμε και μάλιστα ανάγλυφα για την ελευθερία του συνεταιρίζεστε, που είναι ιδιαίτερο πρόβλημα στην περιοχή μας γενικά, αλλά και στην σε επαρχίε μα ειδικότερα και για το μέλλον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτό θα πρέπει σαφώ να εμφανίζεται σαν ένα μόνιμο σημείο που θα πρέπει να μα απασχολεί για την κατάσταση, για τη βελτίωση αυτού του δικαιώματο του συνεταιρίζεστε ε, και μεσονόμων αλλά και από πρακτική πλευράς Ορισμένες παρατηρήσεις σας είναι σημαντικές και θα ήθελα να επιμείνω για το γεγονός ότι στην Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, σε νόσεις προσκαλούν για διάλογο αλλά είναι ε, ψεύτικες ε, μασκαρεμένες οργανώσεις ε, είναι οργανώσεις στην υπηρεσία της απέναντι πλευράς ε, και θα πρέπει να κάνω και λογοπαίγνιο στα γαλλικά, σερβίλ και σιβίλ, μεν που υπηρετούν και οι άλλοι που εξυπηρετούν. Εδώ λοιπόν. Θα πρέπει να σας δείξω και ποιες δικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν όσοι ε, υπερασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσπαθούν να συνεταιριστούν, να συνεργαστούν και δυσκολίες πολλές ε, που εμφανίζονται και είναι κάτι το παστική σημασία ε, να μπορούμε επίσης να έχουμε χρήματα και έχει σημασία η δήλωση των εθνών να αντιμετωπίζουμε τρομερές δυσκολίες σε Αιγύπτο, την Ισία και Αλγερία και μάλιστα τώρα πρόσφατα πριν από δέκα μέρες η, Ευρωπαϊ... Αλγερίνη Ένωση γυναικείων δικαιωμάτων δεν μπορούσε να λάβει τα χρήματα που ήθελαν ε, να μας βοηθήσουν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ακόμα κάτι εδώ ε, θα πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται περισσότερη άμεση στήριξή μας και στα πλαίσια αυτά χρειάζεται να μπορούμε να ενεργήσουμε καλύτερα και στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών. Εδώ ολοκληρώνω, ολοκληρώνω σύντομα κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας της υποεπιτροπή σας ακριβώς ε, εδώ για τα κατεπήγοντα μέτρα και τα ε, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για φροντίδα, για άσυλο και στη Ιώτα, το λατινικό, τα εδάφια 2 και 3 για τις κατεπήγωσα βοήθεια και να αντικατήσουμε έτσι την έλλειψη μιας ε, κατάλληλη στρατηγική, όπως και στο Ζ, το λατινικό, τις παραγράφους που έχουν να κάνουν ε, με τις ε, γυναίκες υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ ακριβώ όλα αυτά χρειάζεται μια διαφάνεια και αυτή είναι η εισαγωγή έκθεση στη 19 σελίδα του γαλλικού κειμένου, όπως επίσης 25 και 26 εδάφια για την βίζα ε, την έκτακτη και 29, 30, 31 εδάφια για την κοινή εκπροσώπηση αυτών ε, και το σύστημα προειδοποίησης και τη βάση στοιχείων ε, και χρειαζόμαστε περισσότερες διευκρινήσεις ε, για την εφαρμογή αυτών κυρίως όσον αφορά και τον εμπιστικό εμπιστευτικό χαρακτήρα, πάρα πολλές πρωτοβουλίες, προτεραιότητες, διαδικασίες που επιθυμούμε και μάλιστα έντονα να έχουμε και ελπίζουμε όλα αυτά να ισχύσουν πραγματικά και όσο γίνεται πιο γρήγορα ε, να έχουν ένα συστηματικό χαρακτήρα όλα αυτά και να μπορούν να συμμετέχουν όλοι και εμείς ελπίζουμε έτσι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ειδικότερα για αυτό που εσείς αποκαλείτε έλλειψη Καλή εφαρμογή, και μάλιστα το λέτε πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ. Δύο αγορητέ, δύο ομιλητέ, μάλλον η κυρία Σάκε, Σκιώδη Σύρια, εξ ονόματο της ομάδας των φιλελεύθερων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους προσκεκλημένου ευχαριστώ και για το καλό σχέδιο έκθεσης. Με ικανοποιούν και τα σχόλια σχετικά με τις ημερίδες συνειδητοποίησης. Ορισμένα από τα στοιχεία, τα πρόσθετα στοιχεία που θα πρέπει να, στα οποία θα πρέπει να εμβαθύνουμε για τα προγράμματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα περιληφθούν και στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η υπηρεσία εξωτερικής δράσης χρειάζεται μια συνολική και εντελεχής προσέγγιση, διότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν προτεραιότητα και ε, σε ειρηνευτικές ε, δραστηριότητες. Πρέπει λοιπόν να ενταχθούν και στα εφιστάμενα προγράμματα. Ένα νέο στοιχείο που λαμβάνει τώρα περισσότερη δημοσιότητα είναι η διάσταση online δεν έχουμε ακόμα βέβαια αρκετά ανεπτυγμένο οπλοστάσιο για την προστασία της ελευθερίας έκφρασης online, δηλαδή στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συνεργαζόμαστε και με το νέο Επίτροπο για την ψηφιακή ατζέντα της Ευρώπης. Είναι σημαντικό διότι όταν θα έχουμε περισσότερη συνειδητοποίηση του ρόλου που μπορεί να παίξει η επιγραμμική επικοινωνία θα δούμε με ποιο τρόπο μπορεί τότε αυτή να συμβάλλει στο να θράψουμε ταμπού, στο να πλησιάσουμε περισσότερο τις γυναίκες και να τους δώσουμε φωνή και τα λοιπά και να αυξήσουμε επίσης τη συνειδητοποίηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων μας εδώ στην Ευρώπη. Ένα άλλο θέμα το οποίο με απασχολεί είναι η έννοια της αξιοπιστίας. Όταν θέλουμε να μιλούμε και στον υπόλοιπο κόσμο πρέπει να δούμε και με ποιο τρόπο βλέπουν αυτοί τον ρόλο που δίνουμε εμείς στα ανθρώπινα δικαιώματα. Χρειάζεται λοιπόν κάποιο μέσον, κάποιο εργαλείο για να δούμε και πώς γίνεται και η διασύνδεση με τα εγχώρια, με τα εσωτερικά ε, στάνταρτ των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε σήμερα τα σχετικά με το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σημαντικά και για την παρούσα έκθεση, διότι το εμπόριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο, ε, το περίφημο ε, καρότο και το ραβδί, ε, για την περίπτωση και του Ιράν ενδεχομένως. Και είναι σημαντικό να συνεργαστούμε, να, κάνουμε, να διεξαγάγουμε ένα διάλογο και με εκπροσώπους των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτές οι ανταλλαγές απόψεων δεν είναι ίσως τακτικές, ούτε γίνονται αρκετά πυκνά, αλλά είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τις χώρες μέλη, νομίζω γνωρίζουμε όλοι τον εντεταμένο έλεγχο της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας και προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάλι εδώ χρειάζονται ιδιαίτερα benchmark και ένα άλλο στοιχείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ακούστηκε προηγουμένως είναι και το ζήτημα του να χορηγούνται προξενικές θεωρήσεις στους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πρέπει να συζητηθεί λίγο το θέμα. Συζητείται και στις κάτω χώρες αυτή, αυτή τη στιγμή. Έχει και σχέση με το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στις προσπάθειες των χωρών μελών, να τους υπενθυμίσουμε ας πούμε τις δεσμεύσεις τους και διαρωτώμε και ποιο οπλοστάσιο διαθέτουμε έτσι ώστε οι υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων να μην παραμείνουν κάτι στη σφαίρα του φανταστικού για τα οποία μιλάμε δηλαδή αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Με την έννοια αυτή πρέπει να εξετάσουμε και τη συνεκτικότητα των πολιτικών των χωρών μελών, αλλά και την συμπληρωματικότητα, γιατί υπάρχουν και πολιτιστικές διαφορές, όπου οι διάφορες χώρες μέλη δηλαδή δίνουν ίσως βάρος σε διαφορετικά θέματα και λόγω βέβαια εγχώριων ευαισθησιών ε, για ορισμένα πράγματα που έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα λοιπόν συνοχή, συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα. Επίσης να εξετάσουμε και τον διάλογο με την άλλη ακτή του Ατλαντικού και να δούμε και εκεί πώς αντιμετωπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και με ποιες προσπάθειες μπορούμε να συμβάλλουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν, θα χαρώ να εργαστώ ακόμη περισσότερο για να κάνω ακόμα καλύτερη την έκθεση. Ευχαριστώ. Κρίστιαν Πρέντα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω στον Λάσλο Τόκας για το, που είναι ο σκιώδης εισηγητής ε, του ΕΛΚ και δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα. Και στη συνέχεια θα σας πω και κάποια προσωπικά μου σχόλια. Μου ζήτησε λοιπόν ο συνάδελφος να ε, σας παρουσιάσω τις εξής ε, απόψεις. Θα θέλε καταρχάς να συγχαρεί την κυρία Χάουταλα για την έκθεσή της και πιστεύει επίσης ε, ότι πρέπει να χαιρετιστεί η απόφαση της ε, υποεπιτροπής μας ε, να γίνει μια τέτοια έκθεση γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Στόκας, λοιπόν ήθελε να υπενθυμίσει το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες για την προώθηση των αλλαγών στις χώρες ε, από τις οποίες προέρχονται και συνεπώς ε, είναι υποχρέωση των κρατών μελών να τις υπερασπιστούν. Ο συνάδελφός μου θα ήθελε να κάνει κάποιες ε, προτάσεις όσον αφορά το κείμενο, τη διατύπωση. Η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ε, εγχειριδίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αναθεωρήθηκε το 2008. Ο συνάδελφος λοιπόν είναι της απόψεως ότι η συγκήτρια θα έπρεπε καλύτερα να αναφέρεται στο τι πράγματι συμπεριλαμβάνει αυτός ο οδηγός. Δεν πρέπει να υποτιμώνται τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, αντιθέτως πρέπει να τα αξιοποιήσουμε πλήρως. Δεύτερη πρόταση. 16 εκατομμύρια ευρώ περίπου από το 2007 το 2010 διατέθησαν για την προστασία των ε, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό δείχνει σαφέστατα ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Τόκες λοιπόν ε, πιστεύει ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που επιλέγονται για να είναι αποδέκτες τέτοιου είδους φόρων πρέπει να είναι εκείνες που έχουν πραγματική εμπειρία στον τομέα. Η εμπειρία είναι κεφαλαιόδου σημασίας ε, για να μπορέσουμε να ε, καταρτήσουμε προγράμματα βιώσιμα και που πραγματικά θα προστατεύσουν τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο συνάδελφός μου τέλος ε, πιστεύει ότι οι συναντήσεις μεταξύ των υπερασπιστών και των διπλωματών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πρέπει να είναι περισσότερες. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συχνότητα των συναντήσεων αυτών. Οι επαφές αυτές είναι εξαιρετική σημασία για να μπορέσουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα προστασίας ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ε, μου ζήτησε ο συνάδελφος να παρουσιάσω. Και τώρα θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να σας ε, πω και τις δικές μου απόψεις σε σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας του κειμένου που έχει συντάξει η κυρία Χάουταλα. Στην παράγραφο 25 θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε το εξή, ότι οι νέε αντιπροσωπείε των κρατών μελών στι τρίτε χώρε πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα επίγουσας ε, θεώρησης ε, στους υπερασπιστές. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια συγκεκριμένη, μια συγκεκριμένη πολιτική εξέταση των αιτήσεων θεώρησης προς αυτή την κατεύθυνση για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφής η πρότασή μας για ένα τέτοιου είδους ε, σύστημα επίγουσας χορήγησης θεώρησης.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 με ναι, πολλά από αυτά που λέχθηκαν. Το υλικό που έχει κατατεθεί είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα μιλήσω για τα γενικά. Θα αναφερθώ ειδικότερα σε δύο σημαντικούς κατά τη γνώμη μου τομείς. Ασχολούμαστε ιδίως με την προστασία των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό είναι καθήκον μας, όχι μόνο ε, ρεαλιστικό αλλά και ηθικό. Όπου και να βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε. Βλέπω δύο τομείς όπου μπορούν να επιτευχθούν κάποιες πρόοδοι. πρώτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε εξάμεινο αλλάζει η Προεδρία. Παρατηρούμε λοιπόν από ετών τις διάφορες χώρες που αναλαμβάνουν ένα εξάμεινο την Προεδρία να δίνουν διαφορετική σημασία στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προστασία των υπερασπιστών τους. Είναι βέβαια ιδιαίτερα ευτυχής η παρούσα συγκυρία διότι η Ισπανική Προεδρία αποδίδει μεγάλη σημασία στα θέματα αυτό. αυτά. Ωστόσο, χρειάζεται μεγαλύτερη συνέχεια στο έργο αυτό. Είναι καλό που έχουμε λοιπόν τώρα αυτό το μηχανισμό και που είναι υποχρεωτικό να διατηρούνται οι επαφές, να διατηρούνται επαφές δηλαδή των τριών διαδοχικών προεδριών, στο σύνολό τους δηλαδή 18 μήνες. Εγώ πάντως θα ζητήσω τα ανθρώπινα δικαιώματα και η φροντίδα για τους ε, ανθρώπους που δραστηριοποιούνται υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων να ανατίθεται όχι μοναχά ε, υπόθεση, να είναι όχι μοναχά υπόθεση των εξάμενων προθεσμιών έχουμε φτάσει τώρα σε καλύτερο σε καλύτερους ε, καιρούς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε λίγους μήνες θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Διπλωματική Υπηρεσία όπως φαίνεται τουλάχιστον δεν ξέρω εάν θα πρέπει να αποδίδουμε πολύ μεγάλη αξία στον τομέα αυτό βέβαια σε όλες τις χώρες δεν έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ειδικέ μονάδες οι οποίες να ασχολούνται με την προστασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων αλλά και με την χορήγηση βοήθειας σε αυτούς που τα υπερασπίζονται. Όμως αν χάσουμε τώρα την ευκαιρία αυτή φοβούμαι δεν θα μπορέσουμε να επανέλθουμε. Ευχαριστώ, Γκέρενς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ορισμένε παρατηρήσει θα ήθελα να κάνω. Σχετικά με την παράγραφο 6, τέσσερις παρατηρήσεις, ε, αλλά να συγχαρώ την εισηγήτρια για την πολύ καλή ανάλυση και όταν το διαβάζουμε ιδιαίτερα χαιρόμαστε εμείς που είμαστε υπέρ των ε, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην παράγραφο 6, πρώτη παρατήρηση αναφέρεται μια κάποια κριτική στην έκθεση, ίσως να αποτελεί η ύπατη εκπρόσωπο για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, η οποία ήταν αρθρόχων τη της Επιτροπής και η δημιουργία μια κοινή υπηρεσία εξωτερική δράση μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο συγκεκριμένο τομέα. Νομίζω ότι αρετές αυτήν την υπηρεσία αποδίδεται που θα πρέπει ακόμα να αποδείξει ότι τις έχει ε, κάπως καταχρηστικά όλα αυτά να λέμε ότι είπατε εκπρός και λοιπά με τα πλησαβόνα ότι είναι τόσο αποτελεσματική με τόση συνεκτικότητα και λοιπά Έτσι. Ε, μάλλον ε, θα θέλατε να επιμείνετε ότι έχει παρόμοιες δυνατότητες, όχι ότι έχει επιδείξει μέχρι τώρα παρόμοια πράγματα. Μετά, για το δικαίωμα Σύλλου ιδιαίτερα συμπαθητική σαν προσέγγιση και ακόμη κάτι, αλλά μια παρατήρηση να προσθέσω. Να μην... Ε, ε όσες πόλεις δεν είναι ε, δεν συμμετέχουν ε, σε αυτό το δίκτυο δεν θα πρέπει να επεκτηθούν τις ευθύνες τους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει ταυτόχρονα ε, να δούμε ε, ότι δεν είναι μόνο αυτές και οι άλλες να μην κάνουν τίποτα. Θα πρέπει όλοι να λάβουν αυτή την ευθύνη και μήπως θα μπορούσαμε να το προσθέσουμε αυτό για τις ε, πόλεις ασύλο. Και ακόμη κάτι, τρίτη παρατήρηση, αναγνώριση μπορώ να το πω. Και μάλιστα επίσημη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες. Να εξηγήσω τι εννοώ. Σε περιπτώσει σύραξη ένα υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει το θάρρο να εκφράσει την άποψή του, ίσω και αυτό σημαίνει συνήθω αντιμετωπίζει ιδιαίτερε δυσκολίε στη χώρα του. Και αν όμω ε, ανήκουν οι χώρε σε μια διεθνή οργάνωση που έχει τις ίδιες αξίες όπως ακριβώς και ο υπερασπιστή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο οποίο διώκεται στη χώρα του τότε ε, Ποιο είναι το λογικό συμπέρασμα. Εάν αυτός ο Διεθνής Οργανισμός ε, αναγνωρίζει ε, το καθεστώς του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, αυτό ενισχύει και τη θέση του. Ένα παράδειγμα. Σε αφρικανική χώρα, οι υπερασπίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν δυσκολίες να τον γνωρίζουν σαν παρόμοιο και να συνεχίσει ελεύθερο στην δραστηριότητά του αλλά εάν είναι μέλος η χώρα του, της Αφρικανικής Ένωσης, έτσι, κατά την απόψή μου είναι ιδιαίτερα δείχνει καθαρά πως έχει κατάσταση. Λοιπόν, αν λοιπόν ε, ε, αναγνωρίζει αυτές τις βάσεις, αυτές τις αρχές και νομίζω ότι εκείνος θα αναγνωριστεί και σαν υπερασπιστής ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισήμως, λοιπόν, γιατί κανείς δεν θα μπορούσε να είναι αντίθετο με κάτι παρόμοιο. Τέταρτο που θέλω να αναφήξω Γενική φύση παρατήρηση και έχει να κάνει με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπενθυμίσω κάτι τώρα. Ο ε, Ολλανδό Υπουργό Εξωτερικών πριν μερικά χρόνια είχε αναλάβει πρωτοβουλία να συμπεριλάβει ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη για την κατάσταση, μάλιστα στα Ηνωμένα Έθνη, για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Αλλά οι υπόλοιποι δεν συμφώνησαν, ε, δεν πήγαν μαζί του από οικονομική πλευρά στην πλήρωσε η Ολλανδία. Αυτό είναι απέσιο, απαράδεκτο. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη ιδιαίτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσε αναφορέ, τόσε δηλώσει, τόσε συνθήκε, ε, αλλά και πρακτική πλευρά όλα αυτά να εκδηλώνονται συγκεκριμένα, να εκφράζονται έτσι και ακριβώς για την ε, είπατε εκπρόσωπο ε, ε, θα πρέπει εκείνη να λαμβάνει το λόγο και όχι οι υπόλοιποι 27 να μην έχουμε χίλιες δυο διαφορετικές δηλώσεις ε, για είναι κάποιος αντίθετος τότε ίσως θα μπορούσε να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί κατά το όφελός του εκείνος που θα εκδηλώσει την διαφορά. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόσουμε την κατάλληλη μέθοδο ότι ίσως για να κάνουμε κάτι το απλό μπορούμε έτσι να οθηθούμε, να κάνουμε κάτι το καλύτερο και είπα ότι εκπρόσωπος να μπορέσει να έλθει εδώ να μας επισκεφθεί γιατί έχει την αρμοδιότητα την εξουσία αλλά έχει και ειδική ευθύνη για διάλογο με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο εκπρόσωπος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αλήσιο Καπελάνη. Έχετε το λόγο. Θα με ακούν οι συνάδελφοι. Ε, μάλλον κάποιο λάθος υπήρχε με το όνομα και ενδεχομένως και η συνάδελφος από την Ισπανική Προεδρία να θέλει να συμπληρώσει ορισμένα πράγματα. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και επειδή ανέφερε ο κύριος Κόρεν στο θέμα της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών ε, και αυτό μεταφράστηκε σε πολύ συγκεκριμένες κατευθυντήριες ε, ε, γραμμές οι οποίες είναι πολύ ρεαλιστικές γιατί δείχνουν ότι διαχειριζόμαστε μονομένες περιπτώσεις που, η μία, που διαφέρουν μεταξύ τους. Σε σχέση τώρα με το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Χαουτάλα, νομίζω ότι θα έπρεπε να τονίσουμε όλα όσα έχουν ήδη γίνει και ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε επί αυτών. Υπάρχουν ήδη 60 χώρες για τις οποίες έχουμε τοπικές ε, στρατηγικές και η Ισπανική Προεδρία μπορεί και εκείνη να μας πει τι έχει κάνει για την ενημέρωση των στρατηγικών αυτών προκειμένου να υπάρχει πλήρης κάλυψη σε όλες τις χώρες οποίες ε, έχουμε αναλάβει δράση και εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών. Ε, επίσης, η Ισπανική Προεδρία ζήτησε οι διπλωματικές ε, αντιπροσωπείες ε, σε όλες τις χώρες να έχουν ένα σημείο επαφής υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί έτσι θα ήταν ευκολότερα τα πράγματα. Όσον αφορά τώρα την συνεργασία, αναφέρθηκε η Διεθνής ε, Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όπως είπε ο συνάδελφος προηγουμένως 18 ε, εκατομμύρια ε, ευρώ έχουν διατεθεί για την ενίσχυση των υπερασπιστών αυτών σε όλο τον κόσμο. Επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε και ορισμένες πτυχές της δουλειάς των υπερασπιστών, δηλαδή θέλουμε και οι πολιτικές και οι πορεί να συμπεριληφθούν στην ε, ε, στρατηγική που θα παρουσιάσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το συζητήσαμε και χθες. Ε, νομίζω ότι η πρόοδος είναι καλή. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά προτείνουμε να να αυξηθούν ε, τα κονδύλια ε, της ε, Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 3% του συνολικού ποσού σε 4,5% που είναι μια αρκετά σημαντική αύξηση και Βεβαίως, επί της βάσης αυτής θα γίνει και ένας νέος διαγωνισμός ε, για να, ακούσουμε πολύ να λάβουμε πολύ περισσότερες πρόσφορες ε, στο πλαίσιο της ε, ενίσχυσης των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης θα ζητήσουμε από μη κυβερνητικές οργανώσεις να μας ε, βοηθήσουν στο πλαίσιο της αναθεωρημένης στρατηγικής μας. Νομίζω ότι η κυρία Λοχμπάιερ έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, που εργάζονται στον τομέα αυτό, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι η συνοχή μεταξύ των μέσων εσωτερικών και εξωτερικών. Ο κώδικας θεωρήσεων, η εφαρμογή του είναι πάρα πολύ σημαντική στο πλαίσιο αυτό και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο, η δική σας Επιτροπή και η Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι μπορεί όταν οι πόροι ε, μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, να ε, συνδυαστεί με το πρόβλημα της χορήγησης θεωρήσεων. Αυτό όμως είναι κάτι, είναι πραγματική προτεραιότητα να συνδεθούν αυτά τα δύο θέματα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η Ισπανική Προεδρία θα ήθελε να σχολιάσει. Ναι. Πολύ σύντομα, ε, αν και τα περισσότερα ήδη λέχθηκαν, ήθελα μόνο να προσθέσω κάτι σχετικά με το τι κάνει η Ισπανική Προεδρία στα πλαίσια των κατευθυντήρων γραμμών για τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Διότι με τον τρόπο αυτό απαντώ και σε ορισμένα πράγματα που λέχθηκαν στη διάρκεια της συζητήσεως. Οι guidelines αυτές εξασφαλίζουν μια συνέχεια γιατί μας μέμφθηκαν πριν για έλλειψη συνέχειας με την αλλαγή των Προεδριών. Αυτό που προβλέπεται στις guidelines είναι όπως προβλέπετε. Δηλαδή έχουμε ζητήσει από όλες τις πρεσβείες μας αλλά και από τις αντιπροσωπείες να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές. Έχουμε ζητήσει από τις πρεσβείες μας να βάλουν focal points στις ε, αντιπροσωπείες κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόσωπο ανθρώπινο με το οποίο μπορούν να έρθουν σε επαφή οι υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης να τελούνται ετήσιες δύο φορές το χρόνο συναντήσεις με υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο τέλος της κάθε προεδρίας ας πούμε. Απαντώ εδώ στον κύριο που προηγουμένως ότι χρειάζονται περισσότερες συναντήσεις με τους αρμοδίους των πρεσβειών. Δίνεται η δυνατότητα έτσι να αναπτυχθεί και διπλωματική δραστηριότητα επιτόπου να γίνουν πιο γνωστοί οι υπερασπιστέ ανθρώπινων δικαιωμάτων, να υπάρχουν, να λειτουργούν καλύτερα οι επαφέ μαζί του, να ακούγονται οι προτάσει του. Αναφέρομαι επίση στο γεγονό ότι αυτό που και προηγουμένω, ότι η Ισπανική Προεδρία στην Τίνιδα δεν δέχθηκε οι υπερασπιστέ των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Λυπούμε που το άκουσα αυτό. Αλλά είπατε και εσεί ότι στη Μαδρίτη σα δεχθήκαμε θερμά και υπάρχει και εκπροσωπο εκεί της Υποεπιτροπής και στην Ισία υπάρχει ομάδα επαφών για να κάνει τις, ε, για να διεξαγάγει αυτές τις αιτήσει συναντήσεις. Σας ευχαριστώ. Ναι, εσείς. Για να απαντήσω εδώ στο θέμα του παγώματος των κονδυλίων για τις ε, ε, γυναίκε με δημοκρατικά φρονήματα. Τώρα το μάθαμε και με την Τινησία, με τις αρχές είχαμε προβλήματα στο παρελθόν στη χρηματοδότηση ακριβώς ε, με πρωτοβουλία ανθρωπίνων δικαιωμάτων των σχεδίων μας στην Τινησία. Είναι σημαντικό το θέμα, το εξετάζουμε και θα δούμε με τις αρχές. Ευχαριστώ. Καταληκτικά τώρα. Κύριε Χαουτάλα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρατηρήσεις και βλέπω ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης ε, και μπορούμε να είναι ακόμη πιο συγκεκριμένη η έκθεση αυτή. Νομίζω ότι ο εκπρόσωπος ε, της Euromed έθεσε το εξή ζήτημα. Είπατε ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για να ενισχύσουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, είπατε νομίζω ότι οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν πρόσβαση στην ε, δική σας ε, χώρα στις υποδομές που μπορούν να τους βοηθήσουν. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να βελτιωθεί πολύ άμεσα. Επίσης αναφερθήκατε σε προβλήματα ελευθερίας έκφρασης και συνεταιρίζεστε. Εγώ ήμουν στη Λευκορωσία την περασμένη εβδομάδα. Μπορώ να πω ότι η Λευκορωσία είναι μια χώρα στην οποία τα ζητήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ακόμη και οι καλύτερες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, δεν καταχωρούνται πουθενά, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται νομίμως και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα παραβίασης ε, της ε, ε, ελευθερίας του συνεταιρίζεστε. Κοιτάξτε, το πρόβλημα Τη παρενόχληση των οικογενειών των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όταν φεύγουν από μια χώρα δεν ξέρουν τι γίνεται με τις οικογένειές τους, δεν μπορούν να έχουν τη βεβαιότητα ότι θα είναι ασφαλείς. Κύριε Σάρκε, νομίζω ότι αναφερθήκατε στα δικαιώματα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ίντερνετ και την παραβίαση της ελευθερίας ε, της έκφρασης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε ξεχωριστά και έχουμε ήδη δρομολογήσει μια μελέτη για να το εξετάσουμε. Όσον αφορά τώρα τις εμπορικές ε, συμφωνίες, συμφωνίες ε, εγώ έρχομαι από μια χώρα που λέγεται η χώρα της Νόκια. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα της Νόκια με το Ιράν, η μη ιδεολοντολογική συμπεριφορά δηλαδή της ε, διοίκησης της Νόκια σε σχέση με τα συστήματα εποπτείας. Ε, κάποιοι λένε ότι ορισμένοι οργανισμοί τυποποίησης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ζητούν την ύπαρξη τέτοιου ίδιου συστημάτων. Όμως είναι σαφές ότι καμία εταιρεία δεν θα έπρεπε να ε, συναλλάσσεται με καθεστώς το οποίο είναι γνωστό ότι διώκει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και νομίζω ότι αυτή η εταιρεία μεταξύ Nokia, Siemens και του, ε, της επίσημης εταιρείας ε, κινητής τηλεφωνίας, νομίζω ότι λέγεται Iran Telecom στο Ιράν, πραγματικά αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, γίνονται ε, κρατήσεις, γίνονται συλλήψεις, γίνονται μέχρι και δολοφονίες υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα είναι κάτι το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής αλλά και σε διαφορετικό πλαίσιο. Κύριε Πρέντα, σας, σας ευχαριστώ πολύ. Στις δικές σας παρατηρήσεις τονίσατε οι αντιπροσωπείες, ε, οι διπλωματικές ε, αντιπροσωπείες ε, να μπορούν να ζητούν επίγουσα χορήγηση θεώρησης. Υπάρχει όμως μια διαφορά μεταξύ της κατάστασης της χώρες στις οποίες υπάρχουν, υπάρχει το πρόβλημα και του τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες προξενικές κατευθυντήριες γραμμές, ε, ενδεχομένως και στο πλαίσιο της Σέγγεν. Ε, παρόλα αυτά, τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίζονται με πολύ διαφορετικό τρόπο από το ένα κράτος ε, μέλος στο άλλο και ίσως θα έπρεπε να υπάρξει κάποιο συντονισμός. Υπήρχαν και πολλές άλλες παρατηρήσεις ο κύριος Γκέρενς μίλησε για τις πόλεις καταφύγια. Αυτό είναι ένα προαιρετικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή είναι προαιρετική. Η ιδέα είναι ότι οι πόλεις αυτές μπορούν, αν θέλουν, να συμμετέχουν, αλλά δεν θα έπρεπε κανείς να θεωρεί ότι μόνο οι πόλεις ε, καταφύγια είναι αυτές που έχουν ε, υποχρεώσεις ως προς τα ε, δικαιώματα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα λάβω υπόψη όλα αυτά τα σχόλια πριν την παρουσίαση του τελικού, ε, του τελικού σχεδίου έκθεσης. Ε, σας ευχαριστώ πολύ όλους. Πρόεδρος, και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγητριά μας και όλους τους ομιλητές που συμμετείχαν στη συζήτηση. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 16 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι οι ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Έχουμε δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι τη Μπάρμπαρα Λόχ Πίλερ για την Αργεντινή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωβουλευτή που έθεσε το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε παρακολουθήσει κατά τα τελευταία χρόνια το θέμα αυτό και βεβαίως θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την Αργεντινή και το συζητήσαμε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Άμυνας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το συζητήσαμε όμως και με την ε, κοινωνία των πολιτών, με μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπως και με ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους. Λαμβάνουμε υπόψη τις ανησυχίες ε, που εξέφρασε η αξιότιμη Ευρωβουλευτής, αλλά πιστεύουμε ότι η κατάσταση είναι μάλλον θετική. Δεν είναι η μόνη Αργεντινή που είχε στρατιωτικό καθεστώς στη Λατινική Αμερική κατά τα χρόνια αυτά, αλλά είναι βέβαια ε, είναι μία από τις χώρες στις οποίες σημειώνονται πολλές καταχρήσεις ε, και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα ε, σε σχέση με τις δίκες των υπευθύνων τον, ε, του στρατιωτικού καθεστώτος. 150 άτομα θεωρούνται ύποπτοι. 243 υποθέσεις αυτή τη στιγμή είναι εκρεμής. Αυτά είναι τα στοιχεία που λάβαμε από την αντιπροσωπεία μας εχθές. Εκτός από τα αριθμητικά στοιχεία, εκτός από τα δεδομένα αυτά, όλο αυτό, αυτό το θέμα έχει συμβολική σημασία και για τη χώρα και για την ευρύτερη περιοχή και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτά. Για το δεύτερο τμήμα, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προστατεύσει τα ε, θύματα που ακόμη απειλούνται μπορούμε κάτι να κάνουμε, αλλά η κυβέρνηση της Αργεντινής έχει την πρώτη ευθύνη. Εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολύ να ενισχύσουμε τους ε, μη κυβερνητικούς φορείς ε, για να βοηθήσουμε τα θύματα παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρηματοδοτήσαμε πολλά προγράμματα μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κάτι ένα μέσο το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό τελικά, μας έδωσε έναν πολύ ενεργό ρόλο στην όλη διαδικασία. Για παράδειγμα, ομάδα συντονισμού για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πολλοί τοπικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, που παρέχουν ψυχολογική και νομική υποστήριξη ε, στα ε, θύματα. Επίσης, προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην συγκέντρωση αποδυτικών στοιχείων για τις δίκες. Ε, περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ στοιχίζουν τα προγράμματα που ε, αφορούν την ε, περιοχή και θα ήθελα να τονίσω την πρωτοβουλία για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα το μέσο για την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα που μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε πολύ ενεργό ρόλο. Συμπληρωματική ερώτηση από εσά, Μπάρμα. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Αν είναι δυνατόν θα ήθελα να δω τη λίστα αυτή. Καλό είναι που υποστηρίζετε τόσες πολλές πρωτοβουλίες. Ε, βέβαια, λυπούμε γιατί δεν μιλήσατε περισσότερο, διότι βλέπουμε καθαρά, τουλάχιστον τι μου λέει η κοινότητα των μη κρατικών οργανώσεων, ότι αυξάνει η αντίδραση στις ε, δίκες, διότι όσο πλησιάζει κανείς περισσότερο στο να διαπιστώσει ποιοι ήταν οι δράστες, τόσο μεγαλύτερες είναι οι αντιδράσεις ο εκπρόσωπος. Θα σας δώσω τη λίστα βεβαίως αμέσως την έχω μαζί μου. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο μέρος της ερωτήσεώς σας, είναι λεπτή η, βέβαια η ισορροπία. Σημειώνω την ανησυχία σας. Θα επανέλθω, θα συζητήσω με την αντιπροσωπεία. Όμως συνολικά η εκτίμηση είναι θετική σχετικά με το, την αξία που έχει η διαδικασία για ολόκληρη την περιοχή αυτή. Θετική αξία δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Μία ακόμα τελευταία ερώτηση. Πρέντα για το Βιετνάμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομος θα είμαι. Η κατάσταση μας ανησυχεί εκεί στο Βιετνάμ, ε, ανησυχεί την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Τελευταίους μήνες σύλληψη κατά δίκες επρασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, ε, ο έλεγχος ακόμα περισσότερο εδώ, ε, θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή θέση του Βιετνάμ, ενώ η Βιετνάμ έχει την προεδρία φέτος περιοδικά του ΑΣΕΑΝ. Και στο Χανόη ο εκπρόσωπός μας ε, μπόρεσε να εκφράσει την ανησυχία του για αυτό το θέμα στην τελευταία συνάντηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, της 11 Δεκεμβρίου στο Ανόη και επίσης με δημόσια δήλωση 21 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε την καταδίκη σε μακρέ ποινέ φυλάκιση στους υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χανόη και Χοτσιμίχ και ε, επίσης ε, εκπρόσωπος μας στο ΑΝΟ για εμπορικά θέματα ταυτόχρονα έθιξε το θέμα με τον κύριο Ζούινγκ ε, υπουργό αρμόδιο για παρόμοια θέματα εμπορικά του Βιετνάμ και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι το αυταρχικό που εκδηλώνεται και τον Ιανουάριο του 2011 στο συνέδριο του κόμματος ε, στο Βιετνάμ και προσπαθεί ακριβώς να φημώσει τις αντίθετες φωνές το καθεστώς ε, δεν πρόκειται προσπαθεί να ε, σταματήσει τον κόσμο να μην εκφράζεται έτσι και τον Οκτώβριο του 2008 και τον Δεκέμβριο του 2009 Νομίζω ότι όλα αυτά ε, ήταν ωφέλιμα, αυτά που είχαμε πει τότε για μια κάποια πίεση για το Βιετνάμ. Ε, εντάξει, δεν ε, μπορούσα να ενημερώσω, αλλά σχετικά με τα ψηφίσματα αυτά, για να δούμε δύο. Να σας πω ότι η Επιτροπή πραγματικά αποδίδει σημασία ώστε ο διάλογος μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Βιετνάμ να εκφραστεί και μέσω συγκεκριμένων βελτιώσεων έχει να κάνει με την αξιοπιστία και τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας αλλά μέχρι τώρα αυτός ο διάλογος ε, μας χρησιμεύσε ιδιαίτερα για να μπορέσουμε να αναφέρουμε και τις ανησυχίες μας και να δούμε ε, συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας με τη χώρα αυτή, διάφορα παραδείγματα. Εργαζόμαστε με τις αρχές του Βιετνάμ για την ευθύρια του τύπου, ρύθμιση σχετικά με τα μέσα ενημέρωση, Είναι συγκεκριμένο ε, θέμα στα πλαίσια του διαλόγου αυτού. Και ακόμα δεύτερο σημείο που είπαν οι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου, εταιρική σχέση, συνεργασία στα πλαίσια τη διαπραγμάτευση με το Βιετνάμ, η συμφωνία αυτή σίγουρα θα συμπεριλαμβάνει και μία παράγραφο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μία αναφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο επίσης και θεωρούμε ότι με τη συμφωνία αυτή θα μπορέσουμε ακόμα περισσότερο να συνεργαστούμε καλύτερα στον τομέα αυτό. Παρακαλώ προσέξτε κάτι. Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την ΑΣΕΑΝ 15-17 ε, έως 17 Μαρτίου θα είναι στο Ανόη θα αποτελέσει ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να θίξει το θέμα αυτό με τις αρχές του Βιετνάμ, να εκφράσει την απόψή του για το θέμα ε, και εξοδότησε τον πρόεδρο κ. Λάγκεν η Επιτροπή μάλλον τον ενημέρωσε συγγνώμη, για την κατάσταση αυτά και σας ευχαριστώ. Κάτι συμπληρωματικό σαν ερώτηση έχετε? Όχι, απλά και μόνο να σας ευχαριστήσω για την απάντησή σας, τίποτα άλλο. Εγώ ε, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πρέντα που έθεσε το θέμα. Εγώ νομίζω ότι είναι δείγμα αυτό της αυξανόμενης οικονομικής επιρροής της Κίνας σε άλλες χώρες και βλέπουμε ξαφνικά μια αλλαγή στάσεως στο Βιετνάμ. Η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία σχέσεων με τις χώρες ΑΣΕΑΝ παρακολουθεί τα θέματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 17 Μαρτίου, στις 3 το απόγευμα. Ίσως να υπάρξει ένα πρόβλημα για τις 7 Απριλίου. Η πρόεδρος ευχαριστεί τους Γερμινείς.